και όλοι όσοι ενδιαφέρεστε και τις εργασίες μας όχι μόνο στη συγκεκριμένη αίθουσα αλλά και αλλού γιατί μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Μπορούν λοιπόν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, καταρχάς. Μπορούμε? Ωραία. Εγκρίνεται. Τώρα, να πούμε μερικά πράγματα για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Έχουμε την τιμή να είναι εδώ μαζί μας ο Ολλανδός Υπουργό Εξωτερικών, ο Μαξίμ Φερχάγεν, για να μας μιλήσει για μια σημαντική έκθεση της Ολλανδικής Κυβέρνησης για την παιδική εργασία. Έχουμε δει λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα, ειδικότερα για την κυβέρνησή σας, ε, κύριε Υπουργέ. Από ό,τι κατάλαβα, το Συμβούλιο θα εγκρίνει τα συμπεράσματά του τον Ιούνιο για το θέμα αυτό και θα δούμε πώς μπορούν τα ευρωπαϊκά όργανα να συμβάλλουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Με ενημέρωσαν ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1999 άρχισε το ενδιαφέρον σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χαιρόμαστε όλους ιδιαίτερος που είστε εδώ μαζί μας. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο. Thank you. Um, thank you, Mrs. Uh, President. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Χαουτάλα. Χαίρομαι όλους ιδιαίτερος που είμαι εδώ στην ε, συνεδρίασή σας και όπως ε, είπατε κι εσείς ε, μου φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις για το 1999 ήμουν αναπληρωματικό μέλος της ε, Επιτροπής σας ε, και για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι η Επιτροπή σας είναι ακόμη τόσο δραστήρια. Άρχισε λοιπόν εδώ η συμμετοχή μου στο θέμα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειές σας, ειδικά τις δικές σας κυρία Πρόεδρε, αλλά και ε, της ε, Επιτροπής για την προώθηση του προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δίνεται τη, μας δίνεται τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με το πώς μπορεί να προχωρήσει, να προωθήσει τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα του ζητήματος παιδικής εργασίας. Πριν από τρία χρόνια που ανέλαβα καθήκοντα προσπάθησα να είναι το επίκεντρο της Ολλανδικής ε, πολιτικής στα ανθρώπινα δικαιώματα για δύο λόγους. Πρώτον, θεωρώ ότι είναι ηθική υποχρέωση η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο ε, στο κάτω-κάτω πρόκειται για, ανθρώπινα, για δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους ανθρώπους παντού και πάντοτε και συνεπώς ε, είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Και δεύτερον, τα, είναι και δικό μας ε, συμφέρον ε, να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Γιατί συνεισφέρουν ε, στην ανάπτυξη, στην σταθερότητα, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δουλεύει το μικροφωνό μου, ρωτάει μιλητής. Α, ωραία δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί αστάθεια και η Ολλανδία, επειδή είναι σημαντικό εμπορικό εταίρο, επωφελείται από ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω, όταν ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω. Ε, ο ρεαλισμό και το εμπόριο είναι κάτι που μπορεί να συνδυαστεί. Τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως ε, παραβιάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα προωθήσουμε. Κινούμαστε προς ένα σύστημα στο οποίο οι παγκόσμιες και οι περιφερειακές δυνάμεις ε, λειτουργούν ε, από κοινού και υπάρχουν, ανθρώπινες, υπάρχουν αξίες που για μας είναι πολύ σημαντικές και που αποτελούν πολύ σημαντικές προκλήσεις. Οι αναδυόμενε ε, δυνάμεις ε, δεν μοιράζονται πάντοτε του καταπολέμησης παιδικής εργασίας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ως μέλη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εσείς θα εξακολουθείτε να ε, ασκείτε πιέσεις προς την κατεύθυνση αυτή γιατί είναι ένα μέτρο που ε, έχουμε στα χέρια μας για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και η συνθήκη της Λισαβόνας ε, ε, σας δίνει πολύ περισσότερες εξουσίες ως συνομοθέτη. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η απαγόρευση των πολίσεων μπορεί να είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι η δουλειά μου βέβαια, θα έλεγα ότι το ψήφισμα για το θέμα αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ Φερχάγεν ή αλλιώ ε, προφέρεται Φερχάχεν. Είναι από τη νότια Ολλανδία ο Υπουργό Διευκρίνηση, επομένω προφέρεται Φερχάχεν το όνομά του. Δείξατε πόσο δραστήριο μπορεί να είναι ένα κράτος μάλλον ε, στις εξωτερικές του σχέσεις ε, και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν το προβάλλουμε δε σε 27 χώρες μέλη θα έχουμε ε, εξαιρετικές πολιτικές και μάλιστα ελπίζω όλοι να ακολουθήσουν το πραγμαδείγμά σα και να υπάρξει ένα φαινόμενο επιπολασμού και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας υπουργοί να κάνουν το ίδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενθάρρυνσή σας διότι έχουμε κάποια πράγματα εν εξελίξη, έχουμε μια γνωμοδότηση η οποία θα προκύψει από την υποεπιτροπή μας, ο συνάδελφος David Μάρτιν είναι ο αρμόδιος και σχετίζεται με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, πτυχές ε, για ανθρώπινα δικαιώματα και τη ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες και νομίζω ότι είμαστε και προς το τέλος ε, αυτής της γνωμοδότησης να σας επισημάνω εδώ και τον συνάδελφο κύριο ε, Χάουι, το οποίος ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι εισηγητής για θέματα εταιρική κοινωνικής ευθύνης. Επομένως υπάρχουν πολλά πράγματα που μας ενδιαφέρουν και θα συζητήσουμε φυσικά και το ενδεχόμενο ενός ε, ψηφίσματος μαζί με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, όπως μας προτείνατε κι εσείς και ελπίζω να προχωρήσει το θέμα αυτό και να είμαστε κι εμείς δραστήριοι και να έχουμε και πολύ καλά συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Ιούνιο. Να ανοίξω λοιπόν, ε, να ξεκινήσει η συζήτηση. Έχουμε τον κύριο Βέρμαν, την κυρία Όμεν και τον κύριο Χάουιτ που θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριος Μπέρμαν καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας σύντομα, σαφώς, συνέχισε την Ολλανδική παράδοση Τη πρόάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, είμαι και περήφανο που το ακούω, είναι το σωστό και φυσικά προ το συμφέρον μας, πολύ σωστά είπε ο υπουργό. Συμφωνώ απολύτω. Αυτό που διαπιστώνουμε για τα θέματα της παιδικής εργασίας είναι στασιμότητα και λόγω της κρίσεως και ίσως και γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο να ε, δούμε το πιο σκληρό κομμάτι της παιδικής εργασίας, τις χειρότερες μορφές μπορούμε ίσως να τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε, ε, κυρίως στη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου το 70% των εργαζομένων είναι παιδιά. Πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό. Αυτή η στασιμότητα θα είναι και θέμα της διεθνούς διάσκεψης που θα γίνει σήμερα και αύριο στις κατοχώρε. Δυστυχώ εγώ δεν μπορώ να παραστώ, αλλά είναι σαφώς, για όλου μας ε, και με την ακρόαση που κάναμε πριν από δύο εβδομάδες στην Επιτροπή ανάπτυξη, ότι η κοινωνική εταιρική ευθύνη δεν αρκεί. Υπάρχει καλή δημοσιότητα, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, καλή την πίστη κάνουν αυτό που τους αναλογεί, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Και εδώ έχουμε τον Υπουργό που κάνει την πρότασή του, πολύ καλή πρόταση. Ε, δεν υπάρχουν δημόσιε προμήθειε και ενισχύσει για επιχειρήσει που δεν συμπεριφέρονται καλά. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και ούτε επιδοτήσει. Πώς όμως θα γνωρίζουμε ποιες επιχειρήσεις ε, κάνουν το σωστό και ποιες δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, ποιες επιχειρήσεις σέβονται τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι. Δεν είναι απλώς το κάνω το σωστό, είναι το να είμαστε και νομότυποι, βάσει και των νόμων του κάθε κράτους μέλους. Ίσως χρειαζόμαστε αυτό το watchdog, το οποίο ζητάω εδώ και δύο χρόνια, να υπάρχει μια γραμμή άμεσης βοηθείας όπου μπορεί κάποιος να καλέσει και να κατονομάσει και να ε, δώσει στοιχεία για οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση και βλέπω ότι και η Ολλανδική κυβέρνηση το υποστηρίζει. Φυσικά θα μπορούσε να βοηθήσει και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Στον τομέα των εξαγωγών έχουμε μόνο το 5% της παιδικής εργασίας. Επομένως, τα μέτρα για το εμπόριο ναι μεν είναι σημαντικά, αλλά το 95% των παιδιών που εργάζονται δεν είναι στον κλάδο του εμπορίου. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβόλων στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε τα παιδιά να μην χρειάζονται και τα παιδιά ευτυχώς δεν είναι φώκες. Ευτυχώς τα παιδιά χρειάζονται σχολεία ίσως και φώκες να χρειάζονται σχολεία, αλλά τέλο πάντων αυτό είναι αντικείμενο επιστημονική έρευνα. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σε σχολεία και αυτό είναι και ο τομέας όπου όλη η συζήτηση για τη μείωση αναπτυξιακής βοήθειας ε, γίνεται πάρα πολύ άσχημη. Ε, υπάρχουν πολλοί, ακόμα και στην Ολλανδία, που μιλούν για αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια, να συζητάμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες και να λησμονούμε το γεγονός ότι θα χρειαστούν δεκαετίες προκειμένου οι αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να αυτοχρηματοδοτούνται σε θέματα παιδείας και υγείας παρεμπιπτόντως. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο, αλλά προ το παρόν η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να μείνει στο επίπεδο που είναι και να την αυξήσουμε και στο 0,7% ε, που προ το παρόν μόνο οι κάτω χώρε το σέβονται. Νομίζω ότι οι χώρες οι οποίες σκέφτονται να μειώσουν στο ίμιση την αναπτυξιακή βοήθεια δεν λαμβάνουν υπόψη του τα παιδιά ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Μπέρμαν και για την παρατήρησή ε, σας για τη σημασία της αναπτυξιακής βοήθειας. Η κυρία Ομενεράιτε. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εντάσσεται στη γενική συζήτηση των αξιών που συζητάμε στην Ευρώπη και των αξιών που, στις οποίες πιστεύουμε στην Ευρώπη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Χωρίς ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε καν μια σωστή κοινωνία. Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και γι' αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τα ανθρώπινα δικαιώματα από ό,τι κάναμε μέχρι στιγμή. Και αυτό το έκανε ο κύριος Υπουργό όχι μόνο τότε όταν ήταν μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, γιατί θυμάμαι ότι είχατε υποβάλει προ... πολλές προτάσεις τότε. Όταν συζητάμε εδώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίω με κεντρικό θέμα τα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου φαίνεται τον μερό να πούμε ότι όταν δεν την χάνουν σεβασμού τα δικαιώματα αυτά, θα πρέπει εμείς να υψώσουμε τον άστιμό μας. Και θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Υπουργέ, τι πιστεύουν οι συνάδελφοί σας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Εκτός αυτού, όταν συζητάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και παιδιά και παιδική εργασία, πώς θα το λάβουμε υπόψη μας αυτό στη νέα υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων. Το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνουμε. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει ένα ειδικό τμήμα της υπηρεσίας που θα ασχολείται με το θέμα αυτό παγκοσμίως στις πρεσβείες αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά. Αναπτυσσιακή βοήθεια. Και κάτι είπε σχετικό και τάις προηγουμένως. Πώς μπορούμε εμείς ως... Ε, πώς μπορείτε εσείς μάλλον ως Συμβούλιο μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να δράσετε πάνω σε αυτό. Επίσης, εμπορικές συμφωνίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον τομέα αυτό των εμπορικών συμφωνιών. Πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας αυτό το θέμα όμως και να έχουμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες. Και τελευταίο θέμα. Με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της Τουρκίας. Και βλέπω συχνά ότι εκτός από το θέμα της εργασίας των παιδιών που υπάρχει και στην Τουρκία, πολλές φορές υπάρχουν παιδιά στις φυλακές Γιατί παραδείγματο χάρη έριξαν τρει πέτρε. Λοιπόν, θα πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο το θέμα της εργασίας των παιδιών, αλλά και το θέμα των ανηλίκων που πολύ γλίγορα μπαίνουν στις φυλακές. Όχι δικάζονται μόνο, αλλά και καταδικάζονται ή κρατούνται κατά τρόπο που οπωσδήποτε δεν είναι σύμφωνος με την αξιοπρέπεια των παιδιών αυτών. Αυτέ οι παρατηρήσει μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να έχετε μεγάλη επιτυχία στο έργο σα. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Κύριε Υπουργέ, θα ακούσουμε με ενδιαφέρον πώ μπορείτε να προωθήσετε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να ζητήσετε από τι υπηρεσίε να, να εξετάσουν προσεκτικά τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να δείτε τι άλλο μπορεί να γίνει Γιατί ο κύριος κίνδυνος που βλέπω εγώ είναι το θέμα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να έχει μια δομή μέσα στα πλαίσια της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι διπλωμάτες που θα ασχολούνται με τις στρατηγικές για κάθε χώρα εκάστοτε θα αφαιθούν εκτός των ε, ευθυνών αυτών. Και Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Χάουιτ και με βλέπω που και η πρόεδρος. Α, και η κυρία Λόχπιλερ βέβαια. Αλλά είδα ότι και η, η πρόεδρος της αντιπροσωπείας της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά δεν, βλέπω δεν θέλει να πάρει το λόγο. Εντάξει. Η κυρία Λόχπίλερ και μετά ο κύριο Χάουιτ. Σα ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τι συστάσει για την εργασία των παιδιών. Δεν πρόφτασα να μελετήσω όλε αυτέ τι συστάσει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρετε ότι μπορούμε να προετοιμάσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα σχετικό, αν αυτό θα σα βοηθήσει. Έχουμε και στην ημεσία μα διάταξη το θέμα τη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του περασμένου έτου. Και λέγεται ότι θα προετοιμαστεί μια μελέτη για θέματα σχετικά με το εμπόριο ε, και που να σχετίζονται και με την εργασία των παιδιών. Είναι έτοιμη η έκθεση αυτή. Α, ωραία, πολύ ωραία. Μετά λέτε ότι είσαστε υπέρ δεσμευτικών ε, υποχρεώσεων για τις εταιρείε. Είμαι πολύ υπέρ αυτής της ιδέας. Από την άλλη μεριά έχω είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Μπορείτε να μας αναπτύξετε πώς μπορέσατε στην πατρίδα σας να δεσμεύσετε τις εταιρείε να μην ακολουθούν αυτές τις τόσο κακές πρακτικές. Μετά λέτε ότι σε διεθνές επίπεδο ε, δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ε, πρόοδος και ιδίως αναφερόσετε εδώ στις ΗΠΑ. Ποιες είναι οι συστάσεις που έχετε ιδίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτούν, να έχουν μια εντολή για, για διεθνείς διαπραγματεύσεις στην, ε, ε, στο Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, Διεθνής Εργασίας και αλλού. Και τρίτος, μόλις είδα αυτό το δημοσίευμά σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στα πλαίσια της κατορικής πολιτικής. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει αυτό κανένας. Γιατί όταν ε, συζητάμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την εξωτερική πολιτική, είναι πιο εύκολο να το περάσουμε στην πατρίδα μα να να ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει να δούμε πώ σχετίζεται αυτό στα εξωτερικά θέματα, αν το συγκρίνουμε, με την ασφάλεια. Ευχαριστώ, κύριε Σάουιτ. Λειτουργεί το μικρόφωνο. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλησπέρα σα, Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σα. Με ενθαρρύνει μια τέτοια πολύ ισχυρή δήλωση από πλευρά Ολλανδική κυβέρνηση και θα ήθελα να ζητήσω από όλου του συναδέλφου, Ολλανδού και μη, να προσπαθήσουν να προωθήσουν όλα αυτά τα θέματα που μα παρουσιάσατε. Όπω είπε και η πρόεδρο, είμαι εισηγητή εδώ και τρει θητείες για τα θέματα της εταιρική κοινωνική Ευθύνη και θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε σε τρία πράγματα για το θέμα αυτό. Συμφωνώ με αυτό που μόλις είπε η συνάδελφός μου επιχειρήσεις που θα μπορούν να έχουν πιστοποιημένες αλυσίδες ε, παραγωγής ε, ώστε να γνωρίζουμε ότι δεν υπήρξε παιδική εργασία. Είναι κάτι το οποίο ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό εδώ στο Κοινοβούλιο. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Και διαπιστώνω ότι υπάρχει κάποια πρόοδος ε, τουλάχιστον σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, γιατί υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, 20 επιχειρήσεις νομίζω περίπου, έχουν ε, κυρώσει τη σχετική σύμβαση. Θα ήθελα να ρωτήσω, όπως και συνάδελφος, τι πρόοδο έχετε επιτελέσει εσείς με τις Ολλανδικές επιχειρήσεις και τι προβλέπετε ότι θα μπορέσετε να κάνετε στο Συμβούλιο με τις επιχειρήσεις ε, ανα την Ευρωπαϊκή Επικράτεια επί του θέματος. Ε, στο θέμα τώρα των πολιτικών ε, εταιρική ευθύνη ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ολλανδική κυβέρνηση ήταν μία από τι πιο προοδευτικέ κυβερνήσει σε θέματα εταιρική ευθύνη, όχι μόνο σε θέματα που μα παρουσιάσετε σήμερα για την εργασία των παιδιών, αλλά και ε, τις βιώσιμες προμήθειες, ε, την ε, διάθεσή σας να διασυνδέσετε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ με εγγυήσει για τις πιστώσεις εξαγωγών. Είσαστε πρωτοπόροι σε θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους σας στο παρελθόν. Αν υπάρχει μία επίκριση είσαστε στην ε, ομάδα υψηλού επίπεδου για τα θέματα αυτά εδώ και τόσα χρόνια και δεν έχετε καταφέρει να εξάγετε εντό εισαγωγικών αυτέ τις πολιτικές από τη Χάγη στις Βρυξέλλες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και μεγάλη απόσταση. Αυτό είναι θέμα πολιτικού βούληση, όχι μόνο για τη δική σα κυβέρνηση, αλλά για όλε μα τι κυβερνήσει. Αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου δεν έχει βάλει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξή τη και νομίζω ότι ε, η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως δεν ενδιαφερόταν, αλλά νομίζω ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται και ίσως ε, ήγηκε η ώρα να προχωρήσουμε αυτές τις πολιτικές ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σχολιάσετε λίγο λοιπόν ε, τι προσπάθειες κάνετε και τι προσπάθειες θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Έχει κλείσει ο κατάλογος των αγορητών. Νομίζω ότι μπορώ να δώσω το λόγο τώρα στον Υπουργό η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο νομίζω ότι αυξάνεται. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για δεύτερη ή τρίτη γενναία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα θέματα αυτά είναι εγκάρσια και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντάξουμε τα ανθρωπίνα, τα ανθρωπίνα δικαιώματα στις πολιτικές μας και μάλιστα σε πολιτικές ε, τις οποίες μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν ε, να αγγίξουμε σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν, υψωνόταν ένα τεράστιο τείχος. Μπορείτε λοιπόν να απαντήσετε στα ερωτήματα των συναδέλφων. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα σχόλιά τους, για τα καλά τους λόγια και για το γεγονός ότι εκτιμούν τις πολιτικές της Ολλανδικής κυβέρνησης είναι πεπισμένο ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα μόνο αν συνεργαστούμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, Κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο και Κοινοβούλια. Προσβλέπω λοιπόν συνεργασία όχι μόνο στο θέμα αυτό, αλλά και σε άλλους τομείς, ώστε να έχουμε συνδυασμένες προσπάθειες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολό τους. παρά το γεγονό ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εξωτερική πολιτική, όπω είπε η κυρία Λοκπέρ, είναι πολύ πιο εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε από ότι οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί και με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, παραδείγματος χάρη παραβίαση δικαιωμάτων των Ρωμά ε, και η παιδική εργασία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να δούμε. Εγώ Είμαι πεπισμένο ότι και οι κυβερνήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ασχοληθούν με το θέμα, αλλά είμαι πεπισμένο ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει και μπορεί να ασχοληθεί με θέματα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω σε κάποιε ερωτήσει. Όπως επεσήμανε η κυρία Όμεν Ρόιτε στη διάρκεια της παρέμβασής της, Μπορώ να χρησιμοποιήσω και τη μητρική μου γλώσσα. Είμαι ευγνώμων λοιπόν στους διερμηνείς που μπορούν να μας κάνουν τη μετάφραση. Θα αλλάξω λοιπόν στη μητρική μου γλώσσα, στα Ολλανδικά και μετά θα επανέλθω και στην Αγγλική. Προς τον κύριο Τάις Μπέρμαν. Να απαντήσω. Καταρχάς να πω ότι αναγνωρίζω τα όσα κάνετε εσείς ε, στον τομέα αυτό. Έχετε δίκιο όταν ρωτάτε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές ε, της εργασίας των παιδιών. Από τις ε, χειρότερες μορφές, αλλά όχι μόνο αυτές. Αν και εσείς θεωρείτε ότι είναι πολύ πιο εύκολες να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, πιο δύσκολες μορφές, αλλά και επίσης ότι το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο. Δεύτερον, η εξαγωγή προϊόντων τα οποία έχουν παραχθεί με ε, παιδική εργασία, ε, κάτι το οποίο είναι μία υποσυνιστόσα της όλης διαδικασίας. Το να εστιάσουμε στις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, κάτι το οποίο είναι και ο στόχος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία θέλει να πάψει να υπάρχει αυτή η μορφή εργασίας μέχρι το 2016, αποτελεί ουσιαστικά ε, τη γέφυρα προκειμένου να εξαλείψουμε το σύνολο της παιδικής εργασίας, δηλαδή το ευρύτερο πρόβλημα. Συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε το στόχο μας, δηλαδή το γεγονός ότι οποιαδήποτε μορφή παιδικής εργασίας ε, είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, το δικαίωμα στην παιδεία, το δικαίωμα στο να παίζει ένα παιδί και στο δικαίωμα στο να ζει στην παιδική του ηλικία. Μου δίνεται εντύπωση ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μόνο μέσω ενός αμαλγάματος οργάνων. Η ανεπτυξιακή συνεργασία είναι μία δυνατότητα η οποία ίσως επισημάνεται υπερβολικά, αλλά προς το παρόν είναι πιο αποτελεσματική. Μπορούμε να τη διασυνδέσουμε και με κάποιες απειλές. Απειλές, επί παραδείγματι, ε, για εμπορικές παρεμβάσεις. Στην Ινδία είχαμε απολύσεις παιδιών και άνοιγμα σχολείων εντός των εργοστασίων ε, τα οποία μπορούσαν να πηγαίνουν τα παιδιά και αυτή τη στιγμή είχε τελειώσει το μάθημα, ο σχολικός χρόνος, μπορούσαν τα παιδιά να εργαστούν στη συνέχεια. Ανεξαρτατοποιήθηκαν κατά κάποιο τρόπο τα παιδιά από αυτή τη μορφή δραστηριότητας. Υπολογίζεται ότι περίπου 250 εκατομμύρια παιδιά απειλούνται από την παιδική εργασία. Γνωρίζουμε όμως ότι το γεγονός ότι δεν θα μπορεί κάποιος ίσως να εξάγει προϊόντα ε, επειδή έχουν γίνει με παιδική εργασία θα μπορούσε να έχει κάποιες συνέπειες διότι θα υπάρχουν και οικονομικές συνέπειες. Τώρα, οι κάτω χώρες τι κάνουμε εμείς εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν και οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα προϊόν παρήχθη και με παιδική εργασία. Πολλοί καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν τέτοια προϊόντα. Αν υπήρχε επισήμανση λοιπόν ή μάλλον όταν υπάρχει επισήμανση που υποδεικνύει ότι ένα προϊόν έχει παραχθεί και με παιδική εργασία, τότε ο καταναλωτή κατά πάσα πιθανότητα θα προτιμήσει να αγοράσει ένα προϊόν στο οποίο δεν έχει υπάρξει παιδική εργασία για την παραγωγή του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δημιουργηθεί ιδέως ευαισθησία και να κάνουμε και την έκκληση στη διάθεσή μας να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά του κόσμου και όχι μόνο τα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα μπορούν να ζήσουν την παιδική τους ηλικία χωρίς εργασία. Τώρα, επιδοτήσεις ενίσχυση στις εξαγωγές δίνονται από τις δημόσιες αρχές υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δήλωση ότι ο, ο, ετών και ο παραγωγός δεν έχουν χρησιμοποιήσει παιδική εργασία. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε ένα ολόκληρο πακέτο και να ζητούμε ως προϋπόθεση οποιοδήποτε ε, παραγωγός ή προμηθευτής να μην ε, χρησιμοποιεί παιδική εργασία, να μην χρησιμοποιεί παιδιά στην εργασία του. Ε, επιλέχθηκε όμως ένα άλλο σύστημα. Δηλαδή, να δίνεται ευθύνη στις επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει παιδική εργασία, αλλά εάν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα μια τέτοια δήλωση, είναι υποχρεωμένη και η επιχείρηση να επιστρέψει την ενίσχυση, αλλά υπάρχει και ένα επιπλέον πρόστιμο. Οι επιχειρήσεις μπορούν έτσι να αποδείξουν ότι κάνουν κάποια βήματα προκειμένου να εξαλείψουν την παιδική εργασία στην αλυσίδα παραγωγής. Κύριε Όμεν ε, Ρόιτε, ε, η, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι εξωτερικές ε, υπηρεσίες. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αφορούν όλες τις γενικές διευθύνσεις. Η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων ε, και η ομάδα υψηλού επίπεδου, λόγω και των καθηκόντων τους, θα πρέπει να προβάλλουν το έργο τους. Εσείς ρωτήσατε ποιος είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τα θέματα της παιδικής εργασίας. το Υπουργείο Εξωτερικών στην ε, Ολλανδία έχει δημιουργήσει ένα ταμείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο χρησιμοποιείται για την ε, ε, προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτε χώρε όταν δημιουργήθηκε το Ταμείο, μα είπαν ότι θα ήταν βλακώδε να γίνει κάτι τέτοιο και δεν θα μπορούσαν να δαπονεθούν τα κονδύλια από πλευρά πρεβιών. Στην πράξη όμως αυτό που έγινε, οι πρεσβείες απευθείας ήταν αυτές οι οποίες εκπώνησαν τα προγράμματα και ήταν αυτές οι οποίες παρουσίασαν μια σειρά από προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν. Πέρσι διαπιστώσαμε ότι οι πρεσβείες επειδή ακριβώς ήξεραν ότι έχουν στη διάθεσή τους το κονδύλιο αυτό άρχισαν να ζητούν κονδύλια και φαίνεται ότι υπάρχει τάση να ζητείται αύξηση του κονδυλίου και μέχρι τέλους του έτους όλες οι πρεσβείες είναι υποχρεωμένες να οργανώσουν μία διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν αρκεί λοιπόν να υπάρχει ένα ε, κεντρικό πρόσωπο, ένας κεντρικός φορέας ο οποίος δίνει κονδύλια, θα πρέπει να επιστήσουμε και την προσοχή σε όλους όσους ασχολούνται με το θέμα αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε και σχετικές υποχρεώσεις. Περνάει στα αγγλικά τώρα ο υπουργό. Καταρχάς, για να απαντήσω στον κύριο Χάουιτ, στις κάτω χώρες με υποστήριξαν οι οργανώσεις εργαζομένων εργοδοτών. Διότι είπαν ότι καταρχάς συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν οι χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, δεν θέλουμε τα προϊόντα μας να παράγονται από παιδιά τα οποία είναι δουλέμποροι ουσιαστικά, ε, είναι δούλοι ουσιαστικά ε, και ζουν υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες διότι είναι προ το συμφέρον των εργοδοτών να έχουν τέτοια δεσμευτικά μέτρα. Θέλει να υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο. Δεν θέλουν οι άλλε επιχειρήσει να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διότι χρησιμοποιούν την ε, παιδική εργασία και φυσικά είναι φτηνότερο για αυτούς να παράγουν ένα προϊόν. Θέλουν να υπάρχει αντικίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση και συνεργάστηκαν μαζί μου για να ε, υπάρχουν προγράμματα τα οποία σχετίζονται και με τις ε, κυβερνητικές ενισχύσεις. Συνεργαστήκαμε και διαπιστώσαμε ότι όλα είναι δυνατά. Και αφού μπορούμε να το κάνουμε εμείς είναι Προφανέ ότι μπορεί να γίνει και σε άλλες χώρες. Αφού εμείς είμαστε μια εμπορική κατεξοχήν χώρα, Προφανώ μπορεί να γίνει και σε άλλες χώρες. Συνεργαζόμαστε ενεργά με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Ε, συζητούμε και με τα συνδικάτα και με τις επιχειρήσεις, αλλά φυσικά όλα αυτά είναι χρονοβόρα. Ιδίω όταν θέλουμε να έχουμε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, Δυστυχώ δεν είναι τόσο καλά οργανωμένοι όσο στις κάτω χώρες και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Μια τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω για την αναπτυξιακή συνεργασία. Είμαι πεπισμένος ότι το κλειδί για την εξάλληψη της παιδικής εργασίας είναι η αναπτυξιακή συνεργασία. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξοδεύει, δαπανά ένα τεράστιο ποσό για την εκπαίδευση για όλους, την παιδεία για όλους, αλλά νομίζω ότι ο στόχος του να πηγαίνουν όλα τα παιδιά σχολείο θα πρέπει να περιλαμβάνει και πιο συγκεκριμένες ε, δράσεις. Να έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένες δράσεις στοχευμένες ε, στα εργαζόμενα παιδιά. Για παράδειγμα, στην Ινδία δημιουργήθηκαν σχολεία δίπλα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς στους οποίους εργάζονταν παιδιά, δίπλα στα ορυχεία στα οποία εργάζονταν παιδιά, ώστε να βλέπουν η διεισόμαση την εναλλακτική λύση. Και όλο αυτό το διασυνδέσουμε και με ένα πρόγραμμα της συνδικής κυβέρνησης η οποία έδινε δωρεάν γεύματα στο σχολείο. Επομένως υπήρχε κίνητρο να πάει κάποιο σχολείο, να έχει και ένα δωρεάν γεύμα και επομένως ήταν πολύ μεγαλύτερο το κίνητρο και τα παιδιά ε, ίσως το τέλος να πάνε σχολείο. Επίσης πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες να ε, εκπονήσουν προγράμματα για την καταπολέμηση των ε, χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας ε, βάσει και τη Σύμβαση 182 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθηθούν αντίστοιχα προγράμματα. Μία τελευταία παρατήρηση του κυρίου Χάουιτ, ε, ο οποίος ρώτησε πώς αντιμετωπίζει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θέματα αυτά και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε εμείς με αυτούς. Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη στιγμή που η Lady Άστον ανέλαβε το θέμα αυτό, και να σας πω εδώ ότι εγώ συνεργάστηκα μαζί της ε, για να συντάξουμε και την πρόταση η οποία παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο ε, για την ε, παιδική εργασία. Η συνεργασία βελτιώθηκε. Ο, προηγού, ο προκάτοχός της δεν ήταν πολύ θερμός οπαδός του θέματος αυτού. Η Lady Άστον όμως ήταν. Προωθήσαμε λοιπόν τα θέματα τα οποία ήταν ευθύνη της ε, κάθε Άστον. Πρόκειται για ένα συνολικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εμπορικών μέτρων και θεωρούμε ότι είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί το θέμα της παιδικής εργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το προωθήσει βάσει και της έκθεσης που παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Προτείν, υπόσχομαι ε, εκ μέρους και των συναδέλφων ε, τους οποίους ακούσατε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε μαζί σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Ε, υποθέτω ότι πρέπει να βιαστείτε για να πάτε στην επόμενη σας συνάντηση, αλλά θα ήθελα να σας θέσω ένα θέμα που θα ήθελα πολύ να έχω τη συνεργασία σας Το ζήτημα που θα ήθελα να θέσω στο πλε... της ε, παρουσίας σας έχουμε τον διάλογο με το Μεξικό στις 12 ε, Απριλίου πριν από τις 17 ε, Μαΐου στη Μαδρίτη Στη Οαχάκα έγινε στις 27 ε, Απριλίου μια σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων δολοφονήθηκαν ε, σε εκστρατεία αλληλεγγύης ε, με την τοπική κοινότητα αυτοχθόνων στην Οαχάκα και Πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και θα έπρεπε να γίνει συνεπώ στο πλαίσιο τη Συνόδου Κορυφή, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα ατιμορρησία που εξακολουθεί να υφίσταται σε αυτό το τμήμα του κόσμου πάρα πολλέ δολοφονίε χωρί καμία απολύτω έρευνα. Μήπω λοιπόν μπορείτε να κάνετε κάτι για το ζήτημα αυτό. Δεν το λέω αυτό γιατί ένας από τους δύο δολοφονηθέντες ε, ήταν ε, Φινλανδός συμπατριώτης μου με τον οργανισμό, ε, με, το, με την οργάνωση του οποίου συνεργάστηκα πάρα πολύ, αλλά και γιατί είναι ένα ζήτημα στο οποίο φαίνεται ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και μπορούμε να αποδείξουμε ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ενσωματωθεί στην πολιτική μας, την εμπορική για παράδειγμα. Δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια αυτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που ήσασταν εδώ μαζί μας και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα τη ημερήσία διαταξή μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Χάουταλα. Σας διαβεβαιώ ότι στο διάλογό μας με το Μεξικό θα ασχοληθούμε με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σχετική ατιμορρησία σε σχέση βέβαια με τις ε, διάφορες ε, ε, τις παραστρατικές οργανώσεις στην περιοχή και ε, σας ευχαριστώ και πάλι που μας δώσατε, μου δώσατε την ευκαιρία για την ανταλλαγή αυτή απόψε μαζί σας. So any, any break. Χωρίς να διακόψουμε, να συνεχίσουμε στο σημείο 4 τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ε, προσπαθήσω να ε, είμαι πάρα πολύ σύντομη για να μην ε, καθυστερήσουμε με τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Θα έχουμε λοιπόν μία ενημέρωση και κλεισμένων των θυρών για τις και τις τελευταίες διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας στις 2 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι θα γίνει μια κοινή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ρωσίας ε, της, ε, στην, στο πλαίσιο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οπότε θα ήθελα να συνεργαστώ με τις αντιπροσωπείες των χωρών. Έχουμε κάποιες Έχουμε κάποιες επαφές ε, με το Συμβούλιο σε σχέση με την πρόσβαση σε πιστευτικά έγγραφα για το θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια επικοδομητική λύση. Και δεύτερον, το Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, έχει αποφασίσει να αποστείλει μια ad hoc ε, ε, αντιπροσωπεία στην Ουγκάντα για την αναθεώρηση του μηχανισμού του ποινικού δικαστηρίου εκεί και αυτό θα αρχίσει στις 31 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου και η συστατική συνάντηση θα γίνει αυτή την εβδομάδα την Τετάρτη 12 Μαΐου στις 11 η ώρα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα εγκριθεί και ένα ψήφισμα μετά τη δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου για το θέμα αυτό στην ε, Ολομέλεια του Μαΐου. Συνεπώς θα είναι μια πολύ καλή βάση για την αντιπροσωπεία μας για τη βελτίωση της ε, διεθνούς ποινική δικαιοσύνης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πολιτικές ε, ομάδες ότι χρειάζεται γραμματεία όλα τα ονόματα ε, των μελών της αντιπροσωπείας το συντομότερο δυνατό. Η αντιπροσωπεία μας θα μετα μετέβη στις 28 Απριλίου στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών και η υποεπιτροπή μας, ε, η ε, κυρία, Νίζεν, και ο κύριος ε, Κόουιτ πήγαν εκεί, ο κύριος Πρόντι, συγγνώμη, πήγαν εκεί και αναφερθήκαμε και, το, αναφερθήκαμε και στο θέμα του διαλόγου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Μεξικό και τα τραγικά γεγονότα εκεί. Ήθελα επίσης να σας πω για την συνάντησή μου με τον πρέσβη του Μεξικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από διπλωματικής ως πραγματικά την πρέσβη, πρέσβη την πρέσβυρα, γιατί είπε ότι είναι ατύχημα, ε, πραγματικά με σόκαρε αυτή η δήλωση, δεν ήταν καθόλου ατύχημα, ήταν ε, ε, έγκλημα και πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Και τέλος, καλά νέα ε, από την επίσκεψη της είπα της εκπροσώπου ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Άστον μετέβη στην Κίνα και μας και ενημερώθηκαν ότι, ενημερωθήκαμε ότι είχε συναντήσεις ε, με ε, ε, σημαντικούς εκπροσώπους ε, της των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Φαίνεται ότι το άνοιγμα της έκθεσης στη Σαγκάη ε, συνέπεσε με την κράτηση πολλών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σύλληψη και την κράτηση. Πάρα πολλοί βέβαια μετέβησαν στην Κίνα επί τη ευκαιρία των εγγενείων της ε, έκθεσης ε, και δεν έχει δοθεί καμία απολύτως προσοχή ε, σε σχέση με την παραφίαση των δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών στην Σαγκάη. Στις 29 με 30 Απριλίου Είχαμε μία συνάντηση με την οργάνωση Ούμπο και εγώ εξέφρασα την πεποίθησή μου ότι η πρόοδος ε, θα προέλθει από την, ε, το διάλογο μεταξύ των Ουιγούρων ε, και των υπόλοιπων μειονοτήτων προκειμένου να μην υπάρξει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί η κυρία Ανδρική και εγώ αποστήλαμε μία δήλωση σε σχέση με την ε, θανατική καταδίκη στην Ταϊβάν, δεδομένου ότι τέσσερις ε, εκτελέστηκαν ε, γιατί είχαν κρυθεί ένοχοι για ποινικά αδικήματα και επειδή δεν είναι μυστικό βέβαια πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο συνάδελφός μας, ο κύριος Τάνοκ, ε, έχει δημοσίως ε, πει ότι η Ταϊβάν είναι μια όρημη δημοκρατία και έχει δικαίωμα να επιβάλλει την θανατική ποινή. Και επίσης ότι υπάρχουν και άλλες χώρες άλλες δημοκρατίες όπως ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία που εξακολουθούν να επιβάλλουν τη θανατική καταδίκη. Κρίμα που ο κύριο Στάνο δεν εδώ, απλώ σα ενημερώνω. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι είπα ότι εκπρόσωπος ε, κατήγγειλε τις ε, εκτελέσεις. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Φιλιππίνες ε, που τα εξετάσαμε στην τελευταία μας συνάντηση, η Παγκόσμια Οργάνωση κατά του βασανιστηρίου η οποία είναι εξαιρετική στη δουλειά της, μας είπαν ότι ο κύριος Ανουάρ Τιπάση, Φιλιππινέζος, ε, ε, έτυχε ε, πολύ βίαιης ανάκρισης και φαίνεται ότι η αστυνομία τον υποχρέωσε να ομολογήσει εγκλήματα κατά ε, Ισλαμικών ομάδων και επίσης ε, ε, και αυτό και ως αποτέλεσμα εμείς να προβούμε σε δηλώσεις σχετικά με τα ζητήματα των βασανιστήριων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ενδεχομένως κάποιοι από εσά να ήσασταν ε, στην Επιτροπή ε, Εξωτερικών όταν ο κύριος Μπρόκ και ο κύριος Φερκόφστατ ε, παρουσίασαν τις τελευταίες τους προτάσεις και θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις τροπολογίες που υποστηρίζουν. Θέλουν να υπάρξει ένα συγκεκριμένο τμήμα που να αφορά ειδικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην διάδοση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης αλλά δεν θέλω να διαβάσω όλη την τροπολογία. Απλώς αναφέρει ακριβώς, ε, ανεξαρτήτως της μορφής που θα πάρει, να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Απλώς θέλω να σας ενημερώσω, γιατί διαφορετικά μπορεί να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Η δεύτερη τροπολογία που έχουν ε, υποβάλει είναι focal points ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας σε όλες ε, τις ε, αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις διάφορες χώρες. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός ε, Μηχανισμός Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα μέσα τα οποία πρέπει να προετοιμάσουμε και τα οποία πρέπει να υποβάλει η ύπατη εκπρόσωπος ε, ως τμήμα του προγράμματός της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα να σας πω ότι κάποιε μη κυβερνητικέ οργανώσεις που παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση πρότειναν η υποεπιτροπή να καλέσει τις ε, επιτροπές ε, των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων των Ευρωπαϊκών Χωρών, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συζητήσουν ακριβώς αυτό το θέμα. Και θα ήθελα απλώ να το θέσω και σε εσά για να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Είναι πολύ αργά για να το κάνουμε αυτό υπάρχει δυνατότητα αυτής της ε, συνεργασίας μεταξύ ημών και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, βλέπω ότι πρόεδροι αντιπροσωπιών ε, της υποεπιτροπής είναι παρόντες. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς κάτι να ρωτήσει. Ναι, η κυρία Λόχ Μπίλερ υπήρχαν εκτελέσεις ε, πέντε στον αριθμό στο Ιράν σήμερα το πρωί και υποθέτω ότι είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί πριν ε, από την επέτειο των ε, εκλογών στην, τον Ιούνιο. Και είναι κάτι το οποίο είχα, είχαν προαναγγείλει ότι θα κάνουν και συνέβη σήμερα το πρωί. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάουιτ δεν είμαι απόλυτα ενήμερος όσον αφορά αυτή την έκθεση για τις επίθεσεις, αλλά κοιτάζοντας τι έχουν που οι συνάδελφοι και οι δικές σας προτάσεις, δεν ξέρω αν θα ήταν χρήσιμο σήμερα να το συζητήσουμε, πώς μπορούσαμε να σας υποστηρίξουμε. Ε, για τη συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια λέτε. Ναι, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Η ιδέα μου η ιδέα θα ήταν να τονίσουμε ότι χρειάζεται να μιλήσουμε σε επιτροπές, επιτροπές υπεύθυνες για εξωτερικές σχέσεις. Δεν ασχολούμεθα με ε, κοινοβουλικές επιτροπές που ασχολούνται με ε, εσωτερικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. αν συμφωνούν ε, και οι άλλοι, θα μπορούσαμε δηλαδή να καλέσουμε κάποιο μέλη των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων ζήσουμε το θέμα, αλλά πρέπει να το προετοιμάσουμε. Σα ευχαριστώ πάντω. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχουν πολλά, πολύ υπομονετικά άτομα εδώ στην αίθουσα και περιμένουμε να ξαναπετύχουμε να επανέλθουμε στην ημερησία μας διάταξη γιατί προσθέσαμε κάποια θέματα βέβαια. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. Ε, Ευρωπαϊκή πολιτική γυπνίασης προς Ανατολάς και Νότο που εξετάζει την παρουσίαση της έκθεσης προόδου της Κομισιόν στις 28 Απριλίου. Οι κύριες εκθέσεις που θα εξετάσουμε σήμερα είναι μία για την Ουκρανία και μία για την Αίγυπτο. Μπορεί κανείς να πει ξεχάσωρα ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίασης είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πολύ καλό που η υποεπιτροπή μας ασχολείται από την ίδρυσή της το 2007 την διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πολιτική αυτή γυπνίασης. Σήμερα συζητάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει των ετησίων αυτών εκθέσεων. Και μια που έχει αναβληθεί η δημοσίευση, ελπίζουμε ότι η αναλογία αυτή απόψεων θα ληφθεί υπόψη στις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική σας. Θα εξετάσουμε κυρίως, όπως σας είπα, αυτές τις δύο χώρες με κάποια μετά από κάποιες γενικές παρατηρήσεις θα ήθελα να δώσω το λόγο στους προκεκλημένους μας ομιλητές. Καταρχήν, 8 λεπτά παρακαλώ ο καθένας Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Ρουτ Βίσερς να πάρει το λόγο που είναι διευθυντή για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γυπνίεση στην Επιτροπή Συντονισμού αυτής της πολιτικής στην κύρια Ρέλεξ και μετά έχουμε τον κύριο Γκρεγουάρ Τερή από το Ευρωπαϊκό Εθνικό Σώμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα παρουσιάσει ένα έγγραφο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Νότο και στην Ανατολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Βίσας έχει το λόγο πρώτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί, όπως είπατε, πρώτη είχε σαν στόχο να υιοθετήσει η Κομισιόν την αιτήση της ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνία στις τέλη Απριλίου. Για λόγους εσωτερικής πολιτικής της Κομισιόν καθυστερήσαμε κάτι τέτοιο και θα γίνει σε δύο μέρες, δηλαδή την Τετάρτη που μας έρχεται. Οι εκθέσει λοιπόν δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί, θα δημοσιευθούν όμως πολύ γλίγορα. Και τα σχόλια που θα σας κάνω αυτή τη στιγμή και που θα κάνουν και οι συνάδελφοί μου φαντάζομαι από την Κομισιόν βασίζονται κυρίως στο προπαρασκευτικό έργο που κάναμε για να προετοιμάσουμε τις μελέτες αυτές. Η πολιτική γυπνίασης βασίζεται στη δέσμευση Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων τους να προσπίσουν τις αξίες δημοκρατία, ε, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει απόλυτα τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού και πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι σημαντικό τμήμα των προγραμμάτων δράσης στα πλαίσια της πολιτικής γεννήσης που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλους σχεδόν τους εταίρους τους. Τώρα την Τετάρτη που μας έρχεται η Κομισιόν θα εγκρίνει την νέα αυτή ανακοίνωση. Ένα γενικό τμήμα και ειδικές, ε, μια ειδική πελέτη για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής το 2009. Θα αναφέρει η ανακοίνωση αυτή τις εξελίξεις από το 2004-2009. Θα τονίσουμε ότι πολλά έχουν επιτευχθεί Ιδίω στον οικονομικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, η πρόοδος ήταν πιο περιορισμένη όσον αφορά το θέμα του κράτους δικαίου. Και πολλοί από τους εταίρους μας μπόρεσαν να ενταχθούν και να συνυπογράψουν πρωτόκολλα και συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά το πρόβλημα είναι η εφαρμογή αυτών. Επιτέθηκα για πρόοδος στην Αίγυπτο Φερρυπίν, ε, ο ακροτισμός των ε, γεννητικών οργάνων είναι τώρα πια έγκλημα γιατί πρέπει να προσπιστούν τα ανθρωπίνα δικαιώματα των γυναικών. Στην Ουκρανία σημαντική πρόοδος επιτεύχθη για την ελευθερία του τύπου με την κατάργηση των κανόνων τεμνίκη, δηλαδή των συστάσεων της κυβέρνησης, του τι επιτρέπεται να δημοσιευθεί. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμα ικανοποιητικό η πρόοδος στην καταπολέμηση των βασανιστήριων είναι ανεπαρκής. Επίσης υπάρχουν προβλήματα σε πολλές χώρες όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, ιδίως τα ΜΜΕ, η ελευθερία του συναθρίζεται, πολλοί περιορισμοί ε, υπάρχουν ακόμα για τους ε, ηγέτες των, της κοινωνίας των πολιτών και εκείνους που προσπίζουν της πολιτικής ελευθερίας. Η θανατική ποινή εξακολουθεί να ε, επιβάλλεται σε πολλούς ε, γειτονές μας και στην Αίγυπτο. Εκείνοι που ζητούν άσυλο και οι πρόσφυγες δεν την χάνουν τις απόλυτες υποστηρίξεις σε πολλές χώρες ε, γειτονικές. Σε πολλές χώρες ούτε το νομοθετικό πλαίσιο για τις εκλογές, ούτε ο τρόπος οργάνωσης των εκλογών είναι σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα. Από την άλλη μεριά, ε, πρόσφατες εκλογές σε γειτονίες μας ήταν δίκαιες και σωστές, όπως παραδείγματος χάνει φέτος στην Ουκρανία. Σε γενικές γραμμές, η Κομισιόν πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας να βελτιωθεί η καλή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά όλα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι και η βάση για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει προσεκτικά να εξολογήσουμε την πρόοδο, να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και βάσει αυτών να αναπτυχθούν οι σχέσεις μας με τους εταίρους μας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γυτνίασης. Ξέρω ότι μπορούμε να βασιστούμε στην υποστήριξη της Υποεπιτροπής και προσβλέπουμε στη σημερινή συζήτηση που θα μας βοηθήσει να τηλευκάνουμε καλύτερα τα πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μεγάλους εταίρους μας, στην Ουκρανία και την Αίγυπτο, όπου υπάρχουν εδώ πιο ειδικευμένοι και ικανοί συνάδελφοι να σας τα παρουσιάσουν στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίσσας, λέει πρόεδρος μου με τα πολύ ειλικρινά σας σχόλια για την κατάσταση και με χαρά μας θα συνεργαστούμε μαζί σας για τη βελτίωση της κατάστασης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Γκρεγκουάρ Τερί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γαλλικά με την άδειά σας. Εδώ και ένα μήνα η FIDH είχε το ε, το συνέδριό του κάθε τρία χρόνια. γιατί αυτό στο Εριβάν στην Αρμενία, όπου συνεκάρισε 160 οργανώσεις που είναι εθνικές οργανώσεις προάσπισης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Επίτροπος Φίλε είχε την καλοσύνη να παρέμβει ενώπιον των οργανώσεων αυτών στο Ερυβάν. Στο τέλος της παρουσίασης οργανώσαμε μια μικρή συζήτηση με τις 30 περίπου οργανώσεις μέλος ε, της ε, ζώνης γειτνίας της για να δούμε πώς ανέλυαν την συζήτηση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτνίασης. Το αποτέλεσμα είναι κάτι που θα ήθελα να παρουσιάσω στους εκπροσώπους εδώ, ότι δηλαδή για άλλη μια φορά οι αρχές της πολιτικής γυπνίασης θεωρούνται πάρα πολύ βασικές και οι αρχές και τα μέσα. Όσοι προσπίζουν ανθρώπινα δικαιώματα πιστεύουν ότι αυτή η μεθοδολογία της ευρωπαϊκής πολιτικής γυπνίωσης θα πρέπει να συμβάλλει στη βεστίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες της εν λόγω γυπνίασης. Από την άλλη μεριά όμως αυτές οι οργανώσεις μέλη συμφωνούν απόλυτα ότι τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γενίασης για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσης, ακόμη πιο ενισχυτικό, η ευρωπαϊκή πολιτική, όπως έχει καθοριστεί από κάποια κρατημένη, έχετε αντίθετη με τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η ευρωπαϊκή πολιτική για Υπάρχει λοιπόν ένα συνέστημα δυσαρέσκειας, όχι καινούριο, αλλά όσο πάει και πιο έντονο που βέβαια είναι σε σχέση με τις τεράστιες προσδοκίες που έχουν οι άνθρωποι αυτοί από την ευρωπαϊκή πολιτική και με κάτι άλλο που είναι ανησυχητικό για τα θεσμικά όργανα. Αυτή η ανασχέτιση εμβαθύνεται όσο πάει περισσότερο σε αυτούς που κανονικά είναι οι φυσικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική γυπνίαση. Η ανάλυση της ε, ας και των άλλων είναι ότι για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Πολιτική τη να αποδώσει θα πρέπει τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα να αντιμετωπίσουν το, τη διπλή πρόκληση. Να ξαναφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των πολιτικών που σχετίζονται με τις σχέσεις με τις αμφισόμενες αυτές χώρες και οριζόντια, επίσης σημαντικό, να αυξήσουν το mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην οδηγήσουν σε, να καταστήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ένα κλειστό ε, σώμα απομονωμένα. Δηλαδή στην καταπολέμηση για την παράνομη μετανάστευση, για το, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εμπορική πολιτική και ούτω καθεξής. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες προκλήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι που απασχολεί τις ε, οργανώσεις μέλη μας. Το εξής, ότι η πολιτική γυθνίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ε, αντικατοπτρίζει κατά κάποιο τρόπο την πολιτική διεύρυνση με ίδια μέσα κλπ. Η κύρια διαφορά είναι όμως ότι η πολιτική γυθνίωση δεν προσφέρει την πολιτική ένταξη. Τι λοιπόν το ουσιαστικό θέμα του κατά πόσο μπορεί να κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες αυτές εταίρους. Οι πολλές από τις οποίες δεν έχουν σχεδόν καμία βούληση να προχωρήσουν σε μια μεταρρύθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό κατέδειξε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτνίαση θα μπορούσε να συνοδεύσει τις ε, μεταρρυθμίσεις, δεν οδηγεί όμως στο να δώσει ενάβσματα για τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Παραδείγματος χάρη στο Μαρόκο, Όταν το Μαρόκο υπήρχε μια εσωτερική δυναμική για μεταρρύθμιση, η Ευρωπαϊκή Ένωση το συνόδευσε με πολύ μεγάλη πτυχία. Όταν όμως αυτή η ορμή χάθηκε στο Μαρόκο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσε να δώσει αυτά τα συμπληρωματικά ενάβματα για να μπορέσει να επαναφέρει τον λογικό δυναμισμό. Αυτό που είναι πολύ πιο ενισχυτικό όμως είναι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να εφαρμόσει τις δύο κύριες αρχές της πολιτικής γυτνίασης. Το πρώτον, η αρχή σύμφωνα με την οποία υπάρχει κοινή δέσμευση, όπως είπε ο κ. να προωθηθούν οι αμοιβέ αυτές αξίες, δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, αυτή είναι μια αρχή που βασίζεται στο σχέδιο δράσης που εκφράζει την θεωρητική αυτή βούληση κοινή πρόοδου και από την άλλη μεριά την αρχή της διαφοροποίησης. Δηλαδή ότι η πρόοδος θα εξαρτάται από την πραγματική εφαρμογή των κοινοτικών προτεραιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα ήθελα εδώ να βασιστώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα ενό εγγράφου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα και που κατά τη γνώμη μου είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων που καταδεικνύει αυτή την ασυνέπεια, αν θέλετε, των ε, θεσμικών οργάνων. Το ε, πρόγραμμα για την Τινησία 2008-2013 που υιοθετήκε πριν μερικές εβδομάδες και λέει εδώ η κυβέρνηση αποδίδει η τη θυμασία στην αναγκαιότητα εγγύηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σαν προϋπόθεση μιας δικομακρατικής δημοκρατίας ευρωπαϊκού τύπου. Η σταθερότητα χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσίαση των δομών του κράτους και του κόμματος στα συνδικάτα, στα ΜΜΕ, στην επικοινωνία, στον πολιτισμικά θέματα, Όλα αυτά για να χαρακτηριστεί μια κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εδώ και 10 χρόνια στην Τινησία δεν προχωράει. Και περικά το λέει η Κομισιόν. Στη σημερινή κατάσταση σχέση με την Τινησία, ο κύριος στόχος είναι να ενδυναμωθεί ο πολιτικός διάλογος, ιδίως με προοπτική της εμβάθυνσης των σχέσεων προς ένα πιο προχωρημένο καθεστώς. Και τέλος, η Κομισιόν παραμένει δεσμευμένη με τη χώρα αυτή για να μπορέσει να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις ούτως ώστε αργότερα να προχωρήσει στον εκδημοκρατισμό. Διαβάζοντας αυτό το κείμενο και λέμε Ευρωπαϊ... Ε, κοινοβουλευτική δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου, λέμε αντίο στα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί λένε δημοκρατία είναι ευρωπαϊκού τύπου. Και επίσης εγκαταλείπουμε και την αρχή της διαφοροποίησης. Γιατί λέμε, υποστηρίζουμε την νησία να προχωρήσει προς τον εξεχρονισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία θα ακολουθήσουν αργότερα. Επίσης, στο ίδιο αυτό πρόγραμμα υπάρχει ένα κεφάλαιο που χαρακτηρίζει τα 15 με 20 εκατομμύρια ε, ευρώ που θα δοθούν στην νησία για τον εξυγχρονισμό του δικοστικού συστήματος πώς λέω θα χρησιμοποιηθούν. Και καμία στιγμή όταν ορίζονται οι όροι αυτοί δεν αναφέρεται ούτε ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτε η ανεξαρτησία των δικαστικών. Ενώ εδώ και πολλά πολλά χρόνια ζητάμε ο εξυγχρονισμός του δικαστικού σώματος στην Ισία να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί από την άλλη μεριά αυτό το δικοστικό τμήμα αυτή τη στιγμή είναι και κατασταλτικό σώμα για την κυβέρνηση. Ποιε συστάσει θα ήθελα να δώσω στο Κοινοβούλιο, να αναφέρονται πολύ περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλου του τομεί τη εξωτερική πολιτική και να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίω ο, ο δημοσιονομικό έλεγχο, για να μπορέσουν να προωθηθούν τα θέματα αυτά. Ο δεύτερο μεγάλο άξονα, βιάζομαι εδώ για να το προφτάσω, ε, πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο δεν φτάνεται στο ύψος των περιστάσεων, θα πρέπει να ελέγχεται καλύτερα η έκθεση προόδου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποφάνονται ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις, ε, την πρόοδο που έχει γίνει στις χώρες αυτές. Επίσης, να ασκείται δημοκρατικός έλεγχος όσον αφορά τις σχέσεις Επίσης αυτή τη στιγμή το θέμα της ε, ανάπτυξης ας πούμε, το οποίο δεν λαμβάνεται όπως θα έπρεπε υπόψη. Τελειώνω εδώ και αν έχετε ερωτήσεις στη διάθεσή σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις επικριτικές σας παρατηρήσεις. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Βίσενς και οι άλλοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορέσουν να σχολιάσουν τα όσα μας είπατε. Θα ήθελα τώρα με την άδειά σας να περάσουμε στη συζητήση αναχώρα. Προτείνω να γίνει μία συζήτηση αφού ακούσουμε και τις εκθέσεις των δύο χωρών. Θα ακούσουμε δηλαδή δύο σύντομες παρουσιάσεις, μία για την Ουκρανία και μία για την Αίγυπτο. Αν συμφωνείτε, να ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Ράιχολ Μπρέντερ, ο οποίος είναι αναπληρωτής ε, διευθυντής του Τμήματος Ανατολικής ε, Συνεργασίας να λάβει το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση Ρελέξ. Θα, θα με επιτρέψετε να μιλήσω γερμανικά. Μία σημαντική εισαγωγική παρατήρηση έγινε ήδη από το συνάδελφο Ρουτ Κερβίσες ότι το νομικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη, στα ε, κράτη εταίρους μας έχει βελτιωθεί, αλλά η εφαρμογή των νόμων αυτών δεν έχει βελτιωθεί τόσο πολύ και αυτό ισχύει και για την Ουκρανία. Αυτή είναι η γενική παρατήρηση που θέλω να κάνω εισαγωγικά. Δηλαδή η Ουκρανία επιτέλεσε τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο, αλλά όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του νομικού πλαισίου και των δικαιωμάτων υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα κεντρικά σημεία. Τέσσερα θα αναφέρω, θα μπορούσα να προσθέσω και άλλα, αλλά δεν θέλω να κατακαιρματίσω την ομιλία μου. Το πρώτο, ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα αστυνομικά κρατητήρια και στα, στις φυλακές. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις βασανιστήριων και ομολογιών που επιτυχάνονται μόνο με τον τρόπο αυτό. Υπήρχε ένα τμήμα ε, παρακολούθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Υπουργείο Ιστορικών, το οποίο όμως δυστυχώ έκλεισε αυτή τη στιγμή. Πολύ λυπηρό, κατά τη γνώμη μας. Όσον αφορά τα δικαστήρια, είναι επίσης σημαντικό ότι η όρη κράτηση εκεί είναι καλύτερη από ό,τι στην κράτηση στις, ε, στα αστυνομικά τμήματα, αλλά όχι ακόμα ιδανική. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ένα σημαντικό μέσο για την αποφυγή των ε, βασανιστήριων αυτών είναι τακτικές και μη προαναγγελμένες επισκέψεις ε, των αρμοδίων στις φυλακές και η Ουκρανία πραγματικά ε, υπέγραψε το πρωτόκολλο του Ηνωμένου Εθνών κατά των βασιστηρίων και της απάνθρωπης μεταχείρισης των κρατουμένων. Ε, είναι λοιπόν μέλος του πρωτοκόλλου αυτού, αλλά από την άλλη μεριά δεν ε, έχει εφαρμόσει ακόμα αυτά που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αυτό. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η κατάσταση στην αντιμετώπιση των ε, προσφύγων και των ζητούντων άσυλο. Δεν υπάρχει μια παράδοση θετική για κάτι τέτοιο στην Ουκρανία και σύμφωνα με τις απόψεις του είπα του Επιτρόπου για τα, τους πρόφυζιες του Ηνωμένων Εθνών το σύστημα καταγραφής των προσφύγων είναι ανεπαρκές και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ε, τυχές και μη οργανωμένες δράσεις της αστρονομίας στον τομέα. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις καταπάτησης των βασικών δικαιωμάτων των ε, ζητούντων άσυλο, ιδίως των, ε, της αρχής της μη επιστροφής στην πατρίδα τους εκεί δηλαδή που απειλείται η ελευθερία και η ζωή τους εδώ σε σχέση με την, με την αντιμετώπιση των ζητούντων άσυλο και των προσφύγων υπήρχαν περιπτώσεις βίας κατά των ατόμων αυτών. Θα πρέπει και αυτό να το σημειώσουμε. Περνώ τώρα στο θέμα των διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν επαρκή ένδυγα μέσα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ξέρετε, στην Ουκρανία υπάρχουν πάρα πολλές μειονότητες Οι νομικές δυνατότητες όπως είπαμε δεν είναι αρκετά αναπτυγμένες. Αυτό ξεκινάει από την ε, διδασκαλία στις διάφορες γλώσσες. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά ανάμεσα στις δηλώσεις της ε, κυβέρνηση που θέλει να υποστηρίξει τις μειονότητες και τις εκτελεστικές διατάξεις που αφορούν παραδείγματο χάρη τη χρήση των γλωσσών των μειονοτήτων κατά την ε, εκπαίδευση. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στους ε, Τατάρους από την Κρυμαία, οι οποίοι τέλη της δεκαετίας 80 ε, ε, πήραν την άδεια να επανέλθουν στην Κρυμαία και υπάρχουν τεράστια προβλήματα για την επανένταξη των ανθρώπων αυτών. Ιδίω αυτό που είναι πάρα πολύ προβληματικό είναι το θέμα της γης, δηλαδή πώς θα έχουν πρόσβαση σε ιδιοκτησία γης ή επαναφορά των αρχικών τους δικαιωμάτων. Υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα διακρίσεις ε, και προκαταλήψεις υπάρχουν και έναντι των Ρωμά. Ε, υπάρχει το θέμα ότι αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις ε, αντισημιτισμού και διακρίσεις βάρος σεξουαλικών μειονοτήτων επίσης. Κάποιες εξελίξεις μας κάνουν να ανησυχούμε όσον αφορά το θέμα της ελευθερίας της σκέψεις. Ξέρουμε ότι βέβαια η Ουκρανία έκανε μεγάλη πρόοδο, ιδίω σε σχέση και με την προκαλή Επανάσταση, αλλά στις πρόσφατες εξελίξεις υπάρχουν ανησυχητικές φωνές, υπάρχουν επιθέσεις κατά ε, δημοσιογράφων και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες καθίσταται ε, πολύ πιο δύσκολη για, από τις αρχές. Και επίσης ε, υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα θέματα της τηλεόρασης και της ελευθερίας της ε, έκφρασης εκεί. Αυτά είναι τα βασικά σημεία στο διάλογο μας με την Ουκρανία και θα ήθελα να αναφερθώ στο τι κάνει η Κομισιόν τελικά. Βέβαια, η συμμετοχή της Ουκρανίας την ευρωπαϊκή πολιτική σα είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητάμε ακριβώς αυτά τα θέματα με την Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία ανέλαβε υποχρεώσεις και μέσα στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίασης. Και η πολιτική αυτή γειτονίασης λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε εμά να εξετάσουμε αυτά τα θέματα και να φροντίσουμε να τηρεί η Ουκρανία τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Θα ήθελα εδώ να κλείσω τις δηλώσεις μου αναφερόμενο στα κλίγορα στα πολλά μέσα που έχουμε στα χέρια μας. Μπορώ να το παρουσιάσω και πιο αναλυτικά αν θέλετε. Το κεντρικό θέμα είναι ότι εν τελευταία αναλύση βέβαια η Ουκρανία ίδια είναι εκείνη που θα επιλέξει την άγουσα που θα θέλει να ακολουθήσει. Από δική μας σκοπιά όμως είναι απαραίτητο και στον τομέα του εκδοκρατισμού και σε άλλους τομείς να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις επαρκείς σχέσεις με την Ουκρανία και μέσα στα πλαίσια μιας νέας συμφωνίας που προετοιμάζεται όπως ξέρετε. Τα μέσα που έχουμε για να επιδράσουμε επί της Ουκρανίας είναι καταρχήν ο πολιτικός διάλογος. Έχουμε ένα πολύ καλό έχουν πάρα πολύ καλά μέσα που έχουμε αναπτύξει ε, διάφορες ε, επαφές ε, και σε επίπεδο υπουργών και σε επίπεδο υπαλλήλων και ένα βήμα της εσωτερικής ε, ασφάλειας όπου συζητάμε τα θέματα αυτά. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική και η τεχνική μας υποστήριξη και θα ήθελα να τονίσω ότι στο νέο πλαίσιο προγραμματισμού 2008-2013 η Ουκρανία θα πάρει 570 εκατομμύρια ευρώ για τα χρόνια αυτά και μάλιστα το 20 με 30% του ποσού αυτού δίνονται στη, για την ενδυνάμωση των ε, νομικών μεταρρυθμίσεων. Και θα ήθελα τέλος να αναφέρω ότι πέρα από τα μέσα της Κομισιόν και των ε, κοινοτικών μέσων και τα κράτη-μέλη παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες κρατών μελών για την προώθηση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρέντερ φαίνεται ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούν να συνεισφέρουν το Κοινοβούλιο και η Υποεπιτροπή, ώστε όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας αναφέρατε μπορούν να, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά. Να ακούσουμε τώρα μία ακόμα παρουσίαση για την κατάσταση στην Ουκρανία και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Ρωμάνα Ρωμανόφ από το πρόγραμμα κράτους δικαίου, είναι διευθυντής του προγράμματος από το Ίδρυμα International Arena σας ε, στο Κίεβο. Μπορείτε να μας πείτε και λίγα λόγια για το Ινστιτούτο σας πριν ξεκινήσετε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι συζητάτε το θέμα της Ουκρανίας αυτές τις ακροάσεις ε, εδώ στην Επιτροπή σας. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, διότι δεν συμβαίνει και πολύ συχνά κάτι τέτοιο. Η Ουκρανία άλλωστε δεν είναι και χειρότερη των περιπτώσεων στην ε, περιοχή. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι θα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι γνωστή στην Ουκρανία ως αυτός που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. αν ε, ε, ρωτήσετε ποιο στην Ευρώπη προωθεί τα ανθρωπίνα δικαιώματα στην Ουκρανία, κατά πάσα πιθανότητα η απάντηση θα είναι Συμβούλιο τη Ευρώπη. Είμαι εκπρόσωπο του International Renaissance Foundation, που είναι το ίδρυμα που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Ε, διευθύνω το πρόγραμμα εδώ και 8 χρόνια και Διαχειριζόμαστε περίπου 50 προγράμματα το χρόνο σε θέματα ποινική δικαιοσύνη, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντίστοιχα θέματα να σας αναφέρω τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα και κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί οι τρέχοντες μηχανισμοί υποστήριξης της ανάπτυξης της Ουκρανίας και τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Συμφωνώ ότι η κατάσταση δεν είναι και χειρότερη δυνατή σε σύγκριση με άλλες χώρες εξακολουθούμε να έχουμε πολυφωνία στη δημοκρατία στην Ουκρανία και φυσικά η Ουκρανία κατάφερε να διασφαλίσει για άλλη μια φορά τη δυνατότητά της να διεξάγει ε, δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ε, διάφορες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χώρα και ταυτοχρόνως μπορούμε να πούμε ότι το κύριο μέσο που επηρέασε τη χώρα δεν ήταν η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία, διότι οι θύνοντε τη χώρα αναζητούσαν κάτι διαφορετικό, κάτι πέραν τη ε, πολιτική γειτονία και το πρόγραμμα δράση ποτέ δεν ήταν ένα έγγραφο εξορθολογισμού για την πρόοδο. Οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών έλαβαν πολύ σημαντική υποστήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η υποστήριξη αυτή ποτέ δεν θα πρέπει να συνδέεται και με την υποστήριξη που δίνεται στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να επανεξετάσουμε στο μέλλον. Το να προσφέρει κάποιο υποστήριξη στην κυβέρνηση δεν είναι και η καλύτερη στρατηγική για να μεταρρυθμιστεί μια χώρα όπως η Ουκρανία. Χρειάζονται πολύ περισσότερα και πρέπει να ε, καταβάλουμε πολύ σημαντικότερες προσπάθειες για να αναπτυχθεί η χώρα. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να συνεργάζεται στενότερα με άλλες περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, κυρίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό, διότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, διαθέτει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη και τους μηχανισμούς προκειμένου να επηρεάσει τη χώρα και τα προγράμματα τα οποία υλοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι πάντα απολύτως αποτελεσματικά. Αυτό που προσφέρουν περισσότερο στη χώρα είναι η διεθνής εμπειρογνωμοσύνη και η παιδεία. Δεν αρκούν όμως εάν δεν υπάρχει και η κατάλληλη υποστήριξη για τις ομάδες υποστήριξης στη χώρα. η βοήθεια θα πρέπει να οδηγήσει και σε εθνική ιδιοκτησία και αυτό δεν μπορεί να προκύψει μόνο από πλευράς κυβέρνησης. Τους τελευταίους μήνες ε, τώρα, να δούμε τι έγινε μετά τις εκλογές στην Ουκρανία. Υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποια ήδη αναφέρθηκαν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανησυχούν πάρα πολύ για την αλλαγή της πολιτικής ε, του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο εσωτερικός μηχανισμός παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταργήθηκε ουσιαστικά και ο νεοδιοριστής υπουργός δεν ε, πρόσφερε κάτι ως αντίβαρο. Επιπλέον, τα τελευταία πέντε χρόνια οι Υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικών ε, ήταν πολιτικοί, δεν ήταν ε, στρατιωτικοί. Και πλέον έχουμε πολίτες, ε, υπουργούς ε, σε άλλους τομείς μεν, αλλά στα θέματα της αστυνομίας έχουμε και πάλι υπουργό αρμόδιο, ο οποίος είναι στρατι, στρατιωτικός. Και δυστυχώ δεν υπάρχει και θέμα ισότητα των φύλων στη χώρα. Δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα εκπρόσωπο ε, στο Υπουργικό Συμβούλιο και φυσικά η και αυτή εκφράστηκε και ο, ο Πρωθυπουργό Ζάροφ ε, δήλωσε ότι δεν είναι αρμόδιες οι γυναίκες ε, για να κάνουν μεταρρυθμίσεις στις χώρες. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό. Κάτι το οποίο επίσης είναι ιδιαίτερο συνοχλητικό είναι ότι οι πιο σημαντικές προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη χώρα για την ε, διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και ε, ξαφνικά αρχίσαμε να έχουμε και διαμαρτυρίες από πλευράς εφημερίδων, ε, τηλεοπτικών καναλιών που διαμαρτύρονται για λογοκρισία. Έχουμε δύο κανάλια, το One Plus One και το STB, το οποίο, τα οποία είναι ιδιοκτησία ιδιωτών, Και είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν ε, offshore εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμένουν στο Λονδίνο, στο Μονακό, στη Γενέβη. Αλλά τελικά φαίνεται ότι αυτό που θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικά για αυτούς είναι να έχουν φθηνότερα καύσιμα και όχι ανθρώπινα δικαιώματα και κοινοβουλευτικέ ελευθερίες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να λάβουμε πιο σοβαρά υπόψη μας την Ουκρανία από πλευράς ε, διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Η σε κυβέρνηση μου φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική ε, σε θέματα καλής και χρηστής διακυβέρνησης. Η προηγούμενη κυβέρνηση και ο προηγούμενος πρόεδρος απέτυχαν ακριβώς ε, προς αυτή την πτυχή στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ε, εκπονήθηκαν ε, μια σειρά από εκθέσεις οι οποίες περιλάμβαναν εξαιρετικά ε, σχέδια για την ανάπτυξη, μεταρρύθμιση του δικαστικού, νομική συνδρομή και πολλά άλλα, τα οποία ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να επαναεπιβεβαιωθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις από την κυβέρνηση, τον πρόεδρο και την κυβέρνηση και να μην ξεκινήσουμε εκ νέου με νέες έννοιε. διότι κάτι τέτοιο θα είναι χρονοβόρο, θα χρειαστεί χρόνος για να τι εκπονήσουμε εκ νέου, να έχουμε την κατάλληλη διεθνή εμπειρογνωμοσύνη και από εκεί και πέρα να τι εφαρμόσουμε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνδυαστούν οι προσπάθειες διαφόρων δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στο διάλογο με την Ουκρανία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η Ουκρανία χρειάζεται κατεπηγόντως ε, βοήθεια και στον οικονομικό τομέα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να θεωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη στον οικονομικό τομέα της ε, χώρας ε, πρέπει να είναι και η βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φρονώ λοιπόν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξορθολογήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πολύ συγκεκριμένε προτάσεις. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Και γνωρίζω ότι δεν θα κάνουμε συζήτηση τώρα, θα ακούσουμε πρώτα τα της Αιγύπτου. Είμαι λίγο σε δυσάρεστη θέση, διότι το Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σκληρό απέναντι στη Λευκορωσία. Αλλά το Κοινοβούλιο δεν είναι τόσο σκληρό, ε, ούτε καν ε, διαφοροποιημένο αν θέλετε, ε, με τις υπόλοιπες ανατολικές χώρες. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω αυτό το θέμα, αλλά διαισθάνομαι ότι πρέπει να επανεξετάσουμε και την κατάσταση των άλλων πέντε χρονών της ε, ανατολικής πολιτικής γειτονίας. Να περάσουμε τώρα σε μια αξιολόγηση για μια άλλη χώρα, για την Αίγυπτο πιο συγκεκριμένα. Κάναμε πάρα πολλές επαφές με τους Αιγυπτίους και σε υπουργικό επίπεδο τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει και σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου και προέκυψαν και κάποιες αντιδράσεις ε, από αιγυπτιακής πλευράς, από αιγυπτιακής κυβέρνηση πιο συγκεκριμένα και η Αίγυπτος φυσικά είναι πολύ κοντινός γείτονας και πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τους δύο μιλητές να λάβουν το λόγο και οι δύο για περίπου 8 λεπτά Πρώτον, ο κύριος Τόμας Ντούπλα Ντελμοράλ, ο οποίος είναι διευθυντής της ε, Γενικής Διεύθυνσης F, που είναι η Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Νότιας Μεσογείου και εκπροσωπήσει φυσικά την ε, Γενική Διεύθυνση Ρελέξ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Μόατα Ελφεγέρη ο οποίος είναι ο εκτελεκτικός διευθυντής ε, του Ινστιτούτου του Καΐρου για τις Μελέτες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του EMHRN, ε, υπεύθυνος για το ENP. Μη με ρωτάτε, λέει η Πρόεδρος, τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά. Α, συγγνώμη, το Δίκτυο Ευρωμεσογειακής συνεργασία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ο κύριο Ντούπλα Ντελμοράλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το, σχέδιο δράσης, ε, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης ε, για τα Δίκτυα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, ισχύει από το 2007 και έχει ένα τμήμα που έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις προστασίας και προώθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τακτικό διάλογο με την Αίγυπτο για τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης ε, παρακολουθεί τις ε, μεταρρυθμίσεις, ε, για παράδειγμα... Το Μάρτιο του 2010 υπήρξε μια υποεπιτροπή που ασχολήθηκε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και είχαμε σε αυτή τη συνάντηση πολύ σημαντικό διάλογο με την Αίγυπτο, ανοιχτό, ε, ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και είδαμε μια επικοδομητική προσέγγιση από πλευρά ε, τη Αιγύπτου. Η Αίγυπτο προσφάτω ε, συμμετείχε στην οικουμενική αναθεώρηση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την περιοδική αναθεώρηση και χαιρετίζουμε το γεγονό ότι συμμετείχαν πολλέ οργανώσει κοινωνία των πολιτών 198 συστάσεις από τις 265 έγιναν ε, αποδεκτές. Τον επόμενο μήνα θα απαντήσει στο, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τις ε, υποθέσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εκκρεμούν και την αφορούν. Είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό αυτό και εμεί θέλουμε όλες ε, οι συστάσεις τις οποίες έχει δεχθεί η Αίγυπτος να συζητηθούν στην επόμενη συνάντησή μας. Αυτό είναι ένα ζήτημα της περιοδικής αναθεώρησης που ήταν τμήμα της ημερήσιας διάταξης εδώ και και θα εξακολουθήσει να αποτελεί τμήμα τη. Έχουμε βέβαια χαιρετήσει τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ελευθερία έκφρασης. Ε, ο αυξανόμενος αριθμός ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης ε, και η μείωση των ποινών ε, για τους δημοσιογράφους ανοίγει τη δυνατότητα ενός διαλόγου που είναι απαραίτητος για την δημοκρατική μεταρρύθμιση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ελευθερία του ε, συναθρίζεστε και έχουν δημιουργήσει μάλιστα και πολλές ανησυχίες. Υπάρχουν ε, πολλές ε, οργανώσεις των κοινωνίων, της κοινωνίας των πολιτών, πολλές διαδηλώσεις, οι οποίες όμως ακόμη αντιμετωπίζουν προβλήματα ελευθερίας έκφρασης και θα έπρεπε να ε, περιοριστούν τα προβλήματα αυτά. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σε σχέση με τη συνέχιση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης ε, στην Αίγυπτο και το γεγονός ε, ότι έχει παραταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλέ φορέ ζητήσει από την Αίγυπτο να εγκρίνει έναν αντιτρομοκρατικό νόμο που να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα. Επίση, μα ενδιαφέρει όλο ιδιαίτερο να μάθουμε τι εγγυήσει ε, ε, από, ε, από αυτά που ακούσαμε στις, 5 Μαΐου θα, θα μεταφραστούν όντω σε νομοθεσία σε σχέση με την τρομοκρατία και την αντιμετώπιση τη εμπορία ναρκωτικών. Το θέμα του βασανισμού επίσης εξακολουθεί να υφίσταται. Η, Ευρωπαϊκή, η Αίγυπτος έχει δεσμευθεί ε, για την αναθεώρηση του, ε, της σχετικής νομοθεσίας ε, και επίσης είπε ότι θα καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να γίνει έρευνα για όλους τους ισχυρισμού βασανισμού. Εμεί εκτιμούμε την ύπαρξη ενεργού συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στην Αίγυπτο. Η συμμετοχή στην διαδικασία ε, UPR είχαν, είχε ως αποτέλεσμα ε, μεγαλύτερο άνοιγμα, περισσότερη ελευθερία έκφρασης και ελπίζουμε ότι η τοποποίηση της ε, νομοθεσίας δεν θα περιορίσει την πρόοδο αυτό, αυτή. Ε, η κυβέρνηση έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων που ανήκουν σε θρησκευτικέ μειονότητε, αλλά παραμένουν προβλήματα, όπω για παράδειγμα η νομική βάση για του τόπου λατρεία. Ε, χρειάζεται να, να αναθεωρηθεί, να μεταρρυθμιστεί και εν ώψη των επερχόμενων εκλογών ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την παρατήρηση των εκλογών. Πολλά ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα ε, τον δικαστικό τομέα ε, πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με το κατά πόσο συνάδουν με διεθνή πρότυπα. Η Αίγυπτος μας είπε ότι δεν έχει σκοπό να δεχθεί παρατηρητές Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων οργανισμών στις εκλογές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει στηρίζει την Αίγυπτο στον εκδημοκρατισμό της με οικονομική υποστήριξη. 45 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί ε, στην ε, Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο ε, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 50 εκατομμύρια μέχρι το 2014 για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι τοπικές οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών επίσης λαμβάνουν υποστήριξη μέσω της του οργανισμού ε, εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κάιρο. Επίσης, σε σχέση, με το, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γειτονίας, ε, θεωρείται η βάση για την, ε, τον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου, η ενίσχυση του διαλόγου αυτού ε, είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που έχει ήδη δρομολογηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την Αίγυπτο να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της για τον εκδημοκρατισμό για να μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος σε ζητήματα δημοκρατίας και ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά βέβαια είναι δυνατά για γιατί χρειάζεται τέτοιου είδους πρόοδος ε, και αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζει και η Αιγυπτιακή κυβέρνηση αλλά και η Αιγυπτιακή κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, πρέπει να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση της Αιγύπτου, να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο περαιτέρω δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και προόδων ε, στον, στα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, ο κύριος Ελφεζιέρη έχει το λόγο. Συγγνώμη αν έκανα λάθος την προφορά. Όχι, μια χαρά το είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι... Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μα ε, ως ε, ε, προσώπου των οργανώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και των ακτιβιστών ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για το ψήφισμα του 2008, το οποίο πραγματικά η κοινωνία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, θεώρησε πολύ ευπρόσδεκτο και χρήσιμο στην Αίγυπτο. Υπήρξε κοινωνική και πολιτική αναστάτωση σε σχέση με το καθεστώς. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση, είναι κάτι το καθημερινό για το εκατομμύρια των Αιγυπτίων. Παράλληλα, συγγνώμη λέει η Πρόεδρος, μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση διατηρεί τις δυνατότητες ε, καταστολής κάθε πολιτική συμμετοχής. Η φιλοδοξία συμμετοχής ε, ε, στο ENP ήταν πολύ υψηλέ το 2005, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Και η Αιγυπτιακή κυβέρνηση που είναι εταίρος σας δεν έχει δείξει πραγματική πολιτική βούληση να δεσμευτεί όντως ε, για το σεβασμό των υποχρεώσεων του σχεδίου δράσης. Επίσης, δεν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα, δεν υπάρχει βαθμολόγιο, δεν υπάρχει συνοχή ε, μεταξύ των οικονομικών μέσων της ευρωπαϊκής της πολιτικής γειτονίας ε, και των υποχρεώσεων ε, της ε, ε, Αιγυπτιακής κυβέρνησης. Παρατηρούμε ότι κάθε συνιστόσα λειτουργεί μεμονωμένα, δεν συνεργάζεται με τις άλλες συνιστώσεις, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και πληροφοριών στα διάφορα διμερεί προγράμματα, τα οποία έχουν αποφασιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονία. Επίση, το μέσο αυτό ε, δεν έχει καταφέρει να, δείξει, να επιδείξει ηγεσία στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη Μεσόγειο ε, και ειδικότερα για μια σημαντική χώρα της περιοχής όπως η Αίγυπτο η ε, Αίγυπτος. Το Μάρτιο του 2005 ε, έγινε η πρώτη προσπάθεια και μέχρι τότε η Αίγυπτος έχει κάνει προσπάθειες. Ε, υπήρξε και έκθεση πρόοδου της Επιτροπής το 2008 βάσει της οποίας δεν υπήρξε πρόοδος στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Ο δείκτης οικονομικής και ανάπτυξης της Αιγύπτου δείχνει τις ανεπάρκειες του συστήματος παροχής βασικών υπηρεσιών στην Αίγυπτο. Και αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διερευνήσει άλλα μέσα συνεργασίας με έναν εταίρο ο οποίος δεν θέλει να ε, αντιμετωπίσει τα βασικά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα της χώρας. Έχουμε, γιατί η Αίγυπτος μπορεί να αξιοποιήσει τα ε, μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση, πρέπει να υπάρχει μια ε, ε, σοβαρή συνεργασία και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει τους Αιγυπτίους ε, ή αν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην πρόθεση των στόχων αυτών. Για παράδειγμα, Προσφάτως ε, μάθαμε ότι η πρόοδος για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι ένας βασικός ε, μοχλός για την Αίγυπτο. Χρειαζόμαστε οικονομική υποστήριξη, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί εφιώς αυτή η υποστήριξη για την, ανθρώπινη, για την ανάπτυξη την οικονομική της Αιγύπτου. Γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, σοβαρά μειονεκτήματα γιατί υπάρχει μια πολιτική εξαίρεση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι τη παραβίασης συνήθω δεν, ε, δεν τιμωρούνται. Υπάρχει ατιμορρησία ε, στο εσωτερικό της Αιγύπτου και μάλιστα για πολλέ δεκαετίες. Η, έκτακτη, κατάσταση εκτάκτου ανάγκη ισχύει από το 1981. Μέχρι από τότε ήταν, είναι μια μόνιμη κατάσταση, ελάχιστα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως για παράδειγμα ε, το, δίκαιο της, ε, το δικαίωμα τη προσωπική ελευθερία και το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Και σε πολλές περιπτώσεις βέβαια έχουν, ε, έχουν γίνει δίκες ε, εναντίον τρομοκρατών, αλλά έχουν γίνει και δίκες απλών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι κάτι το συνεχιζόμενο. Η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να δώσει έναν ε, πραγματικό λόγο συνέχισης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι μια τεχνική καταστολής ε, για να εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια ελίτ. Έγινε τροποποίηση του συντάγματος για αντιδρομοκρατικό νόμο, ε, όμως ε, ενδεχομένως ε, να εξακολουθήσει να ισχύει η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι να ισχύσει ο αντιτρομοκρατικός νόμος, δηλαδή για δύο ακόμη χρόνια. Το 1992 κανονικά έπρεπε να είχε, υπάρξει, να είχε εγκριθεί νομοθεσία για τον αντιτρομοκρατικό νόμο και κανονικά οι ειρηνικέ δραστηριότητε και ε, κάποιε δραστηριότητε ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να είναι κολάσιμε. Τα μέτρα αυτά λοιπόν έχουν χρησιμοποιηθεί για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων και είναι κρίμα που το σχέδιο δράσης ε, με την Αίγυπτο και η έκθεση προόδου για την Αίγυπτο ενθαρρύνει την ε, κυβέρνηση ε, να ε, εγκρίνει έναν ε, αντιτρομοκρατικό νόμο όταν αυτός ο αντιτρομοκρατικός νόμος θα συνεχίσει απλώς την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Επίσης το θέμα του βασανισμού είναι κάτι που είναι ρουτίνα στην Αίγυπτο, είναι κάτι το καθημερινό στα αστυνομικά τμήματα, ακόμη και στα, ε, στο, και στα, στα κεντρικά, ε, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της αστυνομίας ε, οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν τη βία εναντίον αμάχων. Για παράδειγμα το 2007 περίπου 8 Αφρικανοί ε, στο Σινά όταν προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα, εκτελέστηκαν. Η Αιγυπτιακή νομοθεσία επιτρέπει τη θανατική καταδίκη και πολλά ε, αδικήματα και επίση υπήρξαν και πολλέ ε, παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα παραβιάσει ε, εναντίον των γυναικών. Έχει βελτιωθεί κάπω η θέση των γυναικών, αλλά παραμένει, εξακολουθεί να, να παραμένουν πολλά προβλήματα. Η πολιτική εξαίρεση, η πολιτική, πολιτικός αποκλεισμός είναι ο σωστός όρος περιγραφής του Αιγυπτιακού πολιτικού συστήματος. Η πολιτική ελίτ μονοπολεί την πολιτική ηγεσία εδώ και χρόνια Υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις ε, συμμετοχής στον δημόσιο βίο μέσω το, της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. Ε, υπάρχουν πολλές, ε, πολλοί περιορισμοί και πολλές καταχρήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας. Το Σύνταγμα περιορίζει επίσης το δικαίωμα του εκλέγεσθε το, ο εκλογικός νόμος επίσης έχει τη δυνατότητα καταστολής πολλών ε, φωνών ε, της αντιπολίτευσης. Έχουμε δει τέτοια περιπτώσεις, για παράδειγμα το 2005 μετά τις ε, εκλογές ε, μέλος της αντιπολίτευσης ε, συνελήφθη και κρατήθηκε και δεν μπορεί να ε, είναι και πάλι υποψήφιο το συγκεκριμένο άτομο ε, λόγω της ε, κατάστασης. Επίσης δεν υπάρχει και δικαίωμα συνεταιρίζεσθε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της κοινωνίας και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ε, ότι η νομοθεσία θα τροποποιηθεί με πολλούς περιορισμούς ε, για την ίδρυση οργανώσεων, ακόμα και για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, ακόμα και για τα φιλανθρωπικά ε, ιδρύματα. Ε, δεν είναι το Υπουργείο υπεύθυνο, είναι η ασφάλεια υπεύθυνη για τέτοιου είδου ζητήματα στην Αίγυπτο. Για παράδειγμα, μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, που ε, επιδοτούνται από διεθνεί οργανισμού έχουν πάρα πολλού περιορισμού στη λειτουργία του. Και μάλιστα σε κάποια εφημερίδα γράφτηκε προσφάτως ότι οι οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σοβαρή απειλή για την κοινωνία και θα έπρεπε να περιορίζονται. Θα είναι πολύ περιοριστική λοιπόν η επερχόμενη νομοθεσία. Και επίσης δεν υπήρχε και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών ε, για την νομοθεσία αυτή. Η διαβούλευση δεν είναι καθόλου επικοδομητική και δεν θα υπάρξουν και σοβαρά αποτέλεσμα από την ε, διαβούλευση που υποτίθεται ότι έκανε η κυβέρνηση της Αιγύπτου. Όσον αφορά λοιπόν ε, την ελευθερία της έκφρασης, εξακολουθεί να περιορίζεται. Τα, οι δημοσιογράφοι ακόμη ε, διώκονται πάρα πολλοί bloggers ε, και ακτιβιστές στο διαδίκτυο έχουν παρενογληθεί και κρατούνται στο πλαίσιο της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Ο Adam Φαντ από το 2008 κρατείται, όπως για παράδειγμα ο Άννα Ραζίρ από την Άνω Αίγυπτο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες συστάσεις που θα θέλαμε εμείς ε, να υποβάλουμε. Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινωνία ε, θα επιφέρει αποτελέσματα στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, επίσης να αναβαθμιστεί η διμερή σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας συγκεκριμένου όρους και προϋποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, ζητούμε μία ε, αποστολή υψηλού επίπεδου για την παρατήρηση των επερχομένων εκλογών να, παρατηρήσουν, να, να παρακολουθήσουν πολύ στενά την κατάσταση στην Αίγυπτο γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία συνδέονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και είναι απαραίτητος παράγοντας για τη σταθεροποίηση της περιοχής. Ευχαριστώ για αυτή την διεξοδικότητα και πολύ συγκεκριμένη έκθεση. Σε περίπτωση που διαρωτάστε ποια είναι η θέση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, αυτή περιλαμβάνεται στα στοιχεία που έχετε στο φάκελό σας. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο και φυσικά στη συνέχεια οι ομιλητές θα μπορέσουν να επανέλθουν, κυρίως αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την ε, πολιτική αυτή προς ε, Ανατολάς και Δυσμάς. ο κύριο Ζήπη, η κυρία Αρνικίνη και στη συνέχεια ο κύριο Χάουιτ και η κυρία Λόμπιλεν. Ο κύριο Ζήπη, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που διαπιστώνουμε εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση γεγονότων. Μιλάμε για την πολιτική γειτονία, αναφερόμαστε σε δύο πολύ σημαντικές χώρες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ουκρανία είναι ένας γείτονας εντός ε, των ευρωπαϊκών ορίων και η Αίγυπτος είναι γείτονας της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτή η διαφεροποίηση δεν επιδρά βέβαια σε κάποια πολιτική μας απόφαση, αλλά είναι γεγονός, διότι ο ένας είναι Ευρωπαίος γείτονας και ο άλλος είναι γείτονας της Ευρώπης. Άκουσα την παρουσίαση της Ουκρανίας, άκουσα και τις παρουσιάσεις για την Αίγυπτο. Νομίζω ότι και οι δύο χώρες αποτελούν τεράστια πρόκληση και για μας. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας καλύτερα. Ο κύριος Ρωμανόφ είπε ότι στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, οι Ουκρανοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι πιο εξοικειωμένοι με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ρόλο που διαδραματίζει και λιγότερο εξοικειωμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβάλλεται τόσο πολύ και υποθέτω ότι και κάποια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λιγότερο γνωστά στους Ουκρανούς. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, αυτό το συμπέρασμα το οποίο προέκυψε από την παρουσίασή σας. όπως και τα άλλα στοιχεία που μας αναφέρατε. Είπατε Ουκρανία, ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται στα μετόπιστα όσον αφορά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά φυσικά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα στοιχείο αρκετά ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι είχαμε δύο γύρους προεδρικών εκλογών έγινε μια σημαντική αλλαγή, δημοκρατική αλλαγή μάλιστα, αλλά πολύ σημαντική, κάτι το οποίο είναι συμβολικό κατά κάποιο τρόπο. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Μπορεί βέβαια η αλλαγή στη συνέχεια να μην μας χαροποιεί και τόσο, μπορεί να το μετανιώσουμε, αλλά νομίζω ότι προς το παρόν η κατάσταση δεν είναι απόλυτα σαφής για τους παρατηρητές. Τον Ιανουάριο είχαμε και ένα ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουκρανία και ένα μεγάλο τμήμα του ψηφίσματος αυτού αφορούσε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ανάλυση μας βασίζεται στο έργο των αντιπροσωπιών μας, τις διάφορες σχετικές αποστολές. και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιοτική αλλαγή και το θέμα της ελευθερίας του τύπου. Ε, αναφερθήκαμε στην προεκλογική εκστρατεία, ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη μας απασχόλησε και επειδή εγώ ήμουν παρατηρητής, ασχολήθηκα και ιδιαίτερα με τη διαφάνεια των εκλογικών διαδικασιών στις εφορευτικές επιτροπές. το έφυξε αυτό το θέμα και οι παρατηρητές άκουσαν με ενδιαφέρον τις απόψεις μου. Υπήρχαν αρκετές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η εκλογική διαδικασία θα είναι διάφανη, κάτι το οποίο επίσης ήταν χωρίς προηγούμενο. Όλες οι χώρες δεν έχουν αντίστοιχα διάφανες διαδικασίες και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το επισημάνουμε αυτό. Τα νομικά δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά ε, επίσης, ανεξάρτητα με τις ε, πολιτικές συμπάθειες ε, που είναι γνωστές ίσως για τα τηλεοπτικά κανάλια της ε, Ουκρανίας. Όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα παρουσίασαν όλους τους σχετικούς υποψηφίους, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για τις προεδρικές αυτές εκλογές. οι αρχές ε, και ο επιχειρηματικός τομέας διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο. Οι επιχειρήσεις έλεγαν ότι θα πρέπει να τηρούνται τα διεθνή πρότυπα. Δεν δόθηκε όμως ε, ίσως ιδέωσα προσοχή σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μένα προσωπικά. Είχαμε κάποιες προσωπικές δηλώσεις ε, από τοπικούς αξιωματικούς στην Ουκρανία και ακούστηκε ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι περίμεναν αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία. Περίμεναν να αλλάξουν οι λειτουργίες και περίμεναν και αλλαγές και στον τρόπο χρηματοδότησης των τοπικών αρχών, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι λίγο πιο ανεξάρτητη από την κεντρική διοίκηση και από τον προπολογισμό αντίστοιχα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προάγουμε την ενότητα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι τεράστια χώρα και διαιρείται σαφώς σε δύο περιοχές και αυτή η ενότητα μπορεί να προαχθεί εάν ε, έχουμε και κατάλληλη ε, διαμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρουμε ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα στην οποία υπερισχύουν οι μειονότητες, κάτι το οποίο φυσικά ενισχύει την κατάσταση που μόλις σας εξέθεσα. Ο κύριος Ρωμάνοφ νομίζω ότι πολύ σωστά Μα υπέδειξε την κατάσταση, διότι μα είπε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, πρέπει να υποστηρίξουμε τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, διότι χωρί την υποστήριξη αυτή δεν θα έχουμε απτά αποτελέσματα και πρόοδο. Αν θέλουμε να έχουμε πλήρη επιτυχία στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε αυτό αποτελεί κανή και αναγκαία συνθήκη. Αν θέλουμε να δούμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες προχωρούν και θέλουμε να δούμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές ε, να αποτελούν ε, τμήμα της καθημερινής λειτουργίας των κυβερνήσεων, τότε όλα αυτά είναι υψίστη σημασία. Όλες αυτές οι πρόοδοι πρέπει να υποστηριχθούν στην Ουκρανία. Ευχαριστώ τον κύριο Τζιμπ και τώρα η κυρία Άνερκιν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους ομιλητές Όλα όσα ακούσαμε ήταν πολύ ενδιαφέροντα για μας. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερως μία από τις δύο χώρες που καλύψαμε σήμερα, η Ουκρανία. Μία ερώτηση προς τον κύριο Ρωμανόβ. Ξέρετε ότι έχουμε μία έκθεση από το Human Rights Watch ε, με ημερομηνία Δεκέμβριο του 2009 και η διατύπωση είναι πολύ σκληρή παρά τις βελτιώσεις λέει, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ ε, αποδυναμωμένα. Οι βασανισμοί και η κακομεταχείριση είναι ακόμα συνήθις πρακτική. Υπάρχουν επιθέσεις ε, μίσους ε, κατά των μειονοτήτων. Υπάρχει αύξηση της επιδημίας HIV-AIDS ε, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το θέμα αυτό. Και υπάρχουν και κάποια στατιστικά στοιχεία. Το κέντρο AIDS ανέφερε πάνω από 13.000 ε, νέες περιπτώσεις ε, φορέων του AIDS ε, το 2009 και η ερώτησή μου προς εσάς είναι κατά πόσον συμφωνείτε με την αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία. Κύριε Μπρέντερ, εσείς αναφερθήκατε στις εθνικές μειονότητες και την ε, παιδεία και την ανάγκη των γλωσσών. Αναφερθήκατε, αναφέρεστε μόνο στους Ουκρανούς Τάταρους ή αναφέρεστε στους μειονότητες εν γέννη. Και θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλιά σας για την κατάσταση των ε, Τάταρων στην Ουκρανία. Και μια ερώτηση προς τους δυο σας ή σε όποιον ε, γνωρίζει περισσότερο μπορεί να απαντήσει για το θέμα αυτό. Ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει ένα πάρα πολύ διάσημο παράδειγμα, την περίπτωση του Γεώργιο Κονγκάτσε, ο οποίος δολοφονήθηκε. Πέρσι τον Ιούλιο ήμασταν εν αναμονή εκλογών και ο Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων ήταν επισήμως ύποπτος ε, για τη διαταγή της δολοφονίας του Γεώργιο Κονγκάτσεφ. Είμαστε στο 2010 Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο στοιχείο για την υπόθεση αυτή. Οι εκλογέ τελείωσαν, έχει εκλογεί νέος πρόεδρος και ξέρετε ότι η υπόθεση αυτή θα εξακολουθήσει να είναι ασαφής και οι ένοχοι θα παραμείνουν ατιμόρυτοι. Thank you, Mrs. Mr. Howitt. Χάουιτ. Πρέπει να φύγω στις 5.30 και δεν θα μπορέσω να ακούσω όλες τις απαντήσεις. Ε, υπάρχει όμως κάποιος εδώ που θα σημειώσει απαντήσεις από τους αδέλφους. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για τις ερωτήσεις που τίθενται για την Ουκρανία. Θα μπορούσε κάποιο από εσά να σχολιάσει την απόφαση της Ουκρανική κυβέρνησης να εφαρμόσει τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση των διακρίσεων επί τη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού το Μάρτιο φέτος. Υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί πλήρως και τι βήματα έχουμε διαπιστώσει ήδη από το Μάρτιο προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Και δεύτερον, Άκουγα πάρα πολύ προσεκτικά, αλλά δεν κατάλαβα κατά πόσον υπάρχουν προτάσεις για συνταγματική μεταρρύθμιση, ε, ώστε και κατά τρόπον μάλιστα ώστε να είναι αποτελεσματικές. Αυτά είναι μία από τις βασικές ε, απαιτήσεις της ε, ε, κοινωνίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ήθελα να ακούσω κάποιες απαντήσεις. Για τα θέματα της Αιγύπτου, όπως ξέρετε κυρία Πρόεδρε, κατόπιν δική σας ε, προσκλήσεως ακούσαμε το δίκτυο της Euromid για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να του ευχαριστήσω και να τους ε, ευχαριστήσω για το έργο τους. Είναι αξιέπαινο. Προσωπικά μετέβη στο Κάιρο προσφάτως και μίλησα και με τοπικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με διευκόλυνε σε αυτή την επίσκεψη. Δύο θέματα για την Αίγυπτο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτον, αν άκουσα και πάλι καλά, έχουμε 45 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δίνονται για βοήθεια για την εκλογική διαδικασία, αλλά δεν μας έχουν καλέσει ως παρατηρητές. Καλά κατάλαβα αν όντω ισχύει κάτι τέτοιο, πραγματικά μου κόβει η ανάσα. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω κατά πόσον αυτή η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, διότι φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν αρκετοί πολίτες από το εκλογικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ε, παραξενευθούν με μια τέτοια απόφαση. Μια δεύτερη ερώτηση. Όταν ήμουν στο Κάιρο και συνάντησα αυτές τις ομάδες ε, οργανώσεων των πολιτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ουσιαστική διαδικασία μεταρρύθμισης. Το ακούσαμε αυτό και από το δίκτυο της Euromed για τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα το απόγευμα. Και πάλι λοιπόν να απευθύνω την ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι προοπτικές ε, θεωρείτε ότι υπάρχουν για μια αυθεντική και ουσιαστική διαδικασία μεταρρύθμισης η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει στην Αίγυπτο και τρίτον και πάλι προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζω για τις εκτελέσεις ε, μεταναστών στα σύνορα. Νομίζω περίπου 90 άτομα δολοφονήθηκαν φέτος και δεν γνωρίζω και τι δράση έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση σε αυτά τα γεγονότα. Θα ήθελα να ακούσω κατά πόσον έγιναν συνεδριάσεις, έγιναν έρευνες, έχουν γίνει ερωτήσεις στους ε, Αιγυπτίους εταίρους μας για τις περιπτώσεις αυτές. Και τέλος, ε, για την Αιγυπτό, θα ήθελα να πω το εξή. Παραδοσιακά είναι καλό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βασικό εταίρο στη διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Πολλέ από τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, πιστεύουν ότι ίσως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι ΗΠΑ Πολιτείες είμαστε διατεθειμένοι να ε, ξεχάσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι μας έχει δοθεί πολιτική υποστήριξη και ε, επειδή ακριβώς έχουμε τύχει αυτής της υποστήριξης στη διαδικασία ειρήνης Μέσης Ανατολής ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα τα δύο αυτά θέματα θα πρέπει να συνδέονται. Είναι βέβαια και ανεξάρτητα μεταξύ των, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να θέσω το ερώτημα και στους δύο μιλωτές. Συμφωνείτε με την ανάλυση αυτή. Διότι νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ακούσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Uh, Ευχαριστώ. Η κυρία Λοχμπίλερ. Uh, okay. Ένα ερώτημα έχω προς τον κύριο Μπρέντερ. Το πάνω και στα γερμανικά. Είχατε πει ότι η Ουκρανία έχει προβλήματα με πρόσφυγες και την ε, μη αποδοχή, μη χωρίς εισόδου στα σύνορα. Ε, είναι χερσαία σύνορα, τα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σύνορα της Ουκρανίας και γι' αυτό δεν έχουμε τόσο ε, τρομακτικές εικόνες όπως από τις θαλάσσιες μεταφορές. Τι γίνεται όμως όσον αφορά με τα θέματα αυτά. Έχει συζητηθεί με τους επιτόπου ανθρώπους, με το Frontex. Η ερώτηση του Ρίτσαρτ Χάουετ επίση, ε, κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής μεταρρύθμισης, προγραμμάτων ουσιαστικής μεταρρύθμισης ε, όσον αφορά στην Αίγυπτο. Και δύο ακόμη ερωτήσεις έχω. Μας είπε ο κύριος ε, Ελφεγγέρη ότι Εξακολουθεί να είναι αρκετά διαδεδομένο ο βασανισμό. Υπήρχε λοιπόν καμία προσπάθεια συμμόρφωση με τι κατευθυντήριε ε, γραμμέ Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, προκειμένου να συμμορφωθεί η Αίγυπτος με αυτές. Επίσης, κατακρίθηκε η έλλειψη συνοχής μεταξύ των διαφόρων μέσων που έχουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε προσκληθεί σε συνεδριάσεις αξιολόγησης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λοχμπίλερ. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε πρώτο το λόγο στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην FIDH, σε γενικές γραμμές για το, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και μετά θα δούμε ε, αναχώρα τις απαντήσεις. Μα δεν υπήρξαν ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις δικές μας παρεμβάσεις. Ε, τα δύο ζητήματα που θα ήθελα να επενθυμίσω και που είναι σημαντικά για μας είναι ο βαθμός ε, στον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι επίκεντρο των συζητήσεων και της αναβάθμισης των σχέσεών μας και με τον Νότο και με τις ανατολικές χώρε και το λέω αυτό στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών και ο βαθμός στον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, έχουν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το άρθρο 21 της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρεται συγκεκριμένα σε μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή με την ε, προώθηση των κοινών αξιών ε, σε όλους τους τομείς εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το λέω ως γενικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βίσελς. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω το εξής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα και στο παρελθόν είναι πολύ ευγνώμων στην υποεπιτροπή σας, ε, αλλά και στι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που προσκαλούνται ε, στην ε, υποεπιτροπή σας και ανταλλάσσουν απόψεις μαζί σας. Γιατί μεταξύ των υψηλών ιδανικών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων μεταξύ των υψηλών δυναμικών ε, των δικών μας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κατάσταση των ανθρώπων στις χώρες αυτές υπάρχει ένας πραγματικό κόσμος και ο βασικός ε, γνώμονάς μα, ε, η βασική μας αρχή είναι ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι έχουμε να κάνουμε με κυρίαρχα κράτη, με κυρίαρχα κράτη που δεν τους ε, υποσχόμαστε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον όχι για την ώρα, και πρέπει συνεπώς ε, να συμπεριφερθούμε με τον απαραίτητο σεβασμό ε, ενώπιον των συγκεκριμένων κρατών. Υπάρχουν μερικές φορές εντάσεις, τις οποίες γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά για να μπορέσουμε να να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Ε, βεβαίως θέλουμε να ακούσουμε την επικοδομητική σας κριτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα ότι είπατε, ότι δεν είπατε ότι, που δεν είπατε ότι θέλετε, ότι δεν μπορείτε να παρέμβετε στα εσωτερικά ζητήματα ε, κρατών. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε ε, επαναλάβει συχνά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους κυρίους Μπρέντερ και Ρωμανόφ για τα ζητήματα αυτά που αφορούν ειδικότερα την Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια ζητήματα ετέθησαν σε σχέση με την Ουκρανία. Θα προσπαθήσω να τα εξετάσω ένα-ένα όσον αφορά την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ήταν σαφές νομίζω στην ε, παρουσίασή μου ότι η κατάσταση ελευθερίας των ε, ε, μέσων ενημέρωσης παρακολουθείται πολύ στενά γιατί υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες είναι ανησυχητικέ και αναφερόμουν σε σωματικές επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, εκφοβισμό και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το γεγονός ε, ότι Ενδεχομένως ε, η πραγματική δολοφόνοι, η ε, του Ογκοκάτσε δεν έχουν ακόμη διωχθεί δεν ξέρουμε και κατά πόσο υπάρχει μία σοβαρή έρευνα προκειμένου οι ε, δολοφόνοι να ε, δικαστούν και να τιμωρηθούν. Όσον αφορά τώρα τις μειονότητες και τους τατάρους της ε, Κρυμαίας, είναι ένα ζήτημα μειονοτήτων που δεν αφορούσε αρχικά την Ουκρανία. Αρχικά βρισκόταν εκτός Ουκρανίας και είναι ένα ζήτημα πολιτιστικό, κοινωνικό και είναι επίσης ένα ζήτημα πολιτικών αποφάσεων ε, και διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων προκειμένου να βοηθήσουμε την, ε, τις μειονότητες αυτές ε, να ενταχθούν στο περιβάλλον τους αυτό. Κάτι το πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι η Ουκρανία μέχρι τώρα δεν έχει εγκρίνει την απαραίτητη νομοθεσία που θα διευκόλυνε τη διαδικασία. Η αναφορά που έκανα στο ζήτημα των γλωσσών και των μειονοτήτων ε, δεν ε, επικεντρωνόταν κυρίως στους δατάρους Κρυμαίας. Ήταν ένα ευρύτερο ε, σχόλιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μειονότητες στην Ουκρανία, δεκάδες και το ζήτημα των γλωσσών παίζει ένα ρόλο σημαντικό σε πολλές περιπτώσεις και δεν είναι ενεργός διάκριση κατά την άποψή μας. Σε μερικές περιπτώσεις η έλλειψη, υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης ε, προκειμένου να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι για να ε, γίνουν σεβαστές ε, οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν σε σχέση με το δικαίωμα των μειονοτήτων να ενταχθούν ακόμη και γλωσσικά. Όσον αφορά το θέμα της ε, σεξουαλικής βίας, θα πρέπει να το ελέγξω και να επανέλθω. Το θέμα των προσφύγων ε, είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό και έχουν πολύ σημαντική θέση οι πρόσφυγες σε αυτό το έγγραφο από τη Human Rights Watch. Ε, είναι γεγονό ότι το συζητήσαμε αυτό το θέμα με την Ουκρανία σε πολλά επίπεδα. Δεν λέω ότι ε, υπήρξε κάτι το πολύ διαφορετικό αλλά μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι αυτό το ζήτημα το διατηρούμε στο πλαίσιο της ε, ημερήσιας διάταξής μας. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας επιβεβαιώσω και έχουμε δεσμευθεί να το παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό στο πλαίσιο των συζητήσεών μας ε, με την Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρουμάνοφ. Ρουμανόφ, συγγνώμη. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν ε, την Ουκρανία, αλλά να ξεκινήσω με την έκθεση του εγγράφου που έχει διανεμηθεί εδώ. Έχετε δύο έγγραφα ε, από την Διεθνή Αμνηστία και από τη Human Rights Watch. Δεν νομίζω ότι αδικατοπτρίζουν τα ζητήματα τα οποία είναι βασικές ανησυχίες των δύο αυτών ε, οργανισμών. Δεν καλύπτουν όλους τους τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ο δηλαδή τα δικαιώματα των προσφύγων, βασανισμός, ρατσισμός ε, ε, αναφέρονται σε αρκετά σημαντικό βαθμό, όπως επίσης και το θέμα του AIDS στη χώρα. Δεν ε, έχω πολλές αμφιβολίες όσον αφορά αυτά τα θέματα και το πόσο σωστά αναφέρονται στο έγγραφο. Ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα που είχε ως ε, αποτέλεσμα πολλές ε, διαμαρτυρίες στην Ουκρανία είναι το θέμα της ε, δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι Ε, πιστεύω ότι πολλοί έχουν όντως ε, ε, καταδικαστεί άνθρωποι που έκαναν εγκλήματα, αλλά όχι υποχρεωτικά αυτοί που ε, τα διέταξαν. Λοιπόν, Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα της ε, ε νοθείας της, ε, των εκλογών και το, του γεγονότος, όλων αυτών των γεγονότων που ακολούθησαν ε, την Πορτοκαλή Επανάσταση. δεν έχουν κριθεί ένοχοι όλοι όσοι θα έπρεπε. Η δίωξη και η αστυνομία εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πολιτική ηγεσία της χώρας και χωρίς να υπάρξει απαραίτητη μεταρρύθμιση του ε, συστήματος δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία ε, της δίωξης των ενόχων και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ε, και δεν μιλάω βέβαια για την ε, προκουρατούρα της ε, Σοβιετική, του σοβιετικού τύπου που έχουμε ακόμη στη χώρα μας. Ε, όσον αφορά το θέμα της, των διακρίσεων, δεν υπάρχει νομοθεσία κατά των διακρίσεων μόνο για το θέμα της ισότητας ανθρώπων και γυναικών. Για όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Αυτό το είπα και στην παρουσίασή μου. Η, έχουμε παρόλα αυτά μια κυβέρνηση στην οποία δεν εκπροσωπούνται οι γυναίκες ε, και υπάρχει σαφής σεξιστική πολιτική. Δεν υπάρχει λοιπόν αποτελεσματικός μηχανισμός εφαρμογής σχετικής νομοθεσίας. Υπάρχουν δύο ενώσεις ε, δικαιωμάτων των γυναικών και θα δούμε, που ασχολούνται με αυτό το θέμα και θα δούμε τώρα ε, πώς θα ασχοληθεί ε, η δικαστική εξουσία με το θέμα αυτό. Ε, όσον αφορά το βασανισμό, είναι γεγονός ότι πάρα πολλές, ε, πάρα υποθέσεις δεν αναφέρονται. Ένα από τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι οι Ουκρανικές αρχές ε, πρέπει να εξετάσουν στο άμεσο μέλλον είναι ότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι ισορροπημένο μετά την τελευταία συνταγματική μεταρρύθμιση. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να μην φτιάξουμε πάλι ε, σε ένα μοντέλο ε, προεδρικό σοβιετικού τύπου που είχαμε στο παρελθόν και ενδεχομένως τελικά σε αυτή την κατάσταση να καταλήξουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι το Συμβούλιο της ε, Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ασχοληθούν με το θέμα αυτό όσον αφορά τα δικαιώματα των προσφύμων. Συγγνώμη, διακόπτη πρόεδρος, δεν έχουμε χρόνο. Είναι ενδεχομένως δικό μου λάθος, δεν λέω ότι φταίτε εσείς. Ναι, το τελευταίο θέμα λέει ο κύριος Ρωμανόφ, ε, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα ε, που αφορούν αυτό το θέμα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση για παράδειγμα. Ακόμη και το καθεστώς του πρόσφυγα δεν προστατεύει το, το κόσμο ε, στην Ουκρανία. Για παράδειγμα, Ρώσος ε, που επισήμως ε, είχε ε, αναγνωριστεί ως πρόσφυγας τελικά εστάλει πίσω στη Ρωσία. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με τα δικαιώματα των προσφύγων στην Ουκρανία. Μάλιστα λέει η Πρόεδρος. Και οι δυο σας αναφερθήκατε στην κατάργηση του τμήματος ε, παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, κάτι το οποίο, ανησυχη... το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Ο κύριος ε, Ντούγκλε Ντελμοράλ ε, μπορεί να αναφερθεί στα της Αιγύπτου. Ναι. Ακούσαμε τους τομείς για τους οποίους η κατάσταση είναι προβληματική. Είναι γεγονός ότι η Αίγυπτος είναι σημαντικός εταίρος λόγω του ρόλου της στον αραβικό κόσμο, του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, το κατά πόσο κάνουμε τα στραβά μάτια στο τι συμβαίνει στην Αίγυπτο, δεν νομίζω. Νομίζω ότι Κάποια από τα πράγματα που ανέφερα στην παρουσίασή μου δείχνουν πόσο ε, προβλήματα που ακούσαμε συζητιούνται. Θα συζητούμε τα προβλήματα. Όλα όσα ανέφερε ο κύριος Ελφετζέρη είναι αντικείμενο συζητήσεων ε, σε ε, συναντήσεις μας ε, στην Υποβιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε επαφές μας με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς, τι θέλουμε να πετύχουμε και πώς θέλουμε να το πετύχουμε. Ένας από τους βασικούς στόχους ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας είναι σύγκληση σε πολλούς τομείς και τη ρυθμιστική ε, σύγκληση και σε οικονομικά ζητήματα σύγκληση. Πιο σημαντικό από όλα όμως είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Εκατέρωθεν της Μεσογείου, εμπροκειμένο. Σε πολύ σημαντικούς τομείς υπάρχει αυτό το χάσμα, στο, στα ποσοστά ανάπτυξης, ε, σε, σε κατακεφαλήνα ΕΠ, ε, σε πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχει βέβαια και το γεγονός του μεγάλου πληθυσμού που ζει στη φτώχεια. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με αξίες ε, που ε, εμείς πρεσβεύουμε ε, εκατέρωθεν της Μεσογείου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα αυτό όσο το δυνατόν καλύτερα και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνο και αν οι εταίροι μας θέλουν να το κάνουμε αυτό. Θέλει λοιπόν η Αίγυπτος να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Έχει σημειώσει πρόοδο ε, στην ανάπτυξη, ε, στη βελτίωση του ΑΕΠ. Βέβαια μπορεί να υπάρχει και ένα φαινόμενο αύξησης της ανισότητας, ε, αλλά συμμετέχουμε στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού τομέα στην Αίγυπτο και άλλων κοινωνικών τομέων. Και αυτό δείχνει ακριβώ πόσο θέλουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτό το χάσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την ε, συνεργασία ε, και σύγκληση στους στόχους μας αυτούς με την Αίγυπτο. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε ε, τον στόχο αυτό με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι τα επιθυμητά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Όσον αφορά τώρα συγκεκριμένα ε, ζητήματα, 45 εκατομμύρια για τις ε, ε, για βοήθεια στις εκλογές όχι γιατί η Αίγυπτος δεν θέλει να κάνουμε κάτι τέτοιο νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το είπα σαφώς όταν έκανα την παρουσίασή μου γιατί η Αίγυπτος δεν θέλει να υπάρξουν παρατηρητές Όσον αφορά τώρα τις ε, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, ε, ναι, πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές πρόπτικες ε, σε διάφορους τομείς και όπως σας είπα η πρόοδος είναι άνηση. Τώρα, το τι έχουμε κάνει για τις δολοφονίες των μεταναστών. Αναφέραμε το θέμα αυτό στο διάλογό μας ε, με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Την ενθαρρύνουμε να, ε, να μην ε, καταφεύγει σε βία σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πυθό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βέβαια η Αιγυπτιακή κυβέρνηση δίνει κάποιους λόγους ε, γιατί τα πράγματα ε, παίρνουν αυτή την τροπή. Προσπαθούμε να τους ακούσουμε, προσπαθούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και το και ο συνάδελφος ε, Βίσελς, έχουμε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα να αντιμετωπίζουμε, έχουμε να κάνουμε με κυρίαρχα κράτη και πρέπει με τις κυβερνήσεις των κυρίαρχων κρατών να συζητήσουμε όσον αφορά το βασανισμό. Αν υπάρχει παρακολούθηση, αν υπάρχει follow-up, ναι, βεβαίως και εδώ και ε, μέσω της αντιπροσωπείας μας ε, προσπαθούμε να θέτουμε το θέμα στους Αιγυπτίους εταίρους μας. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, δεν είναι κάτι που ξεχνάμε. Και πιστεύουμε ότι σε κάποιους τομείς υπάρχουν δεσμεύσεις από πλευράς κυβέρνησης που μας επιτρέπουν την πρόοδο στο μέλλον. Προσπαθούμε λοιπόν ε, σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας να κινηθούμε. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα. Ναι, μπορεί να μην υπάρχει πολύ συνοχή στις διάφορες συνιστώσεις της ε, δουλειάς μας, αλλά αυτό, ε, έτσι είπατε εσείς, αλλά μπορεί να μην είναι αυτός ο λόγος. Ε, οι όροι εφαρμογής και οι συνθήκες εφαρμογής δεν υπάρχουν. Ο κύριος Ελφεζιέρη. Ευχαριστώ. Για τους βασανισμούς. Οι βασανισμοί σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκες ε, και με την έλλειψη μεταρρυθμίσεων. Όπως σας είπα, ε, οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν θα πρέπει να σχετίζονται με συγκεκριμένα μέτρα και ο βασανισμός είναι ένα εξ αυτών. Πρέπει να υπάρχει μια επίσημη εκστρατεία την οποία να ε, προωθεί η κυβέρνηση και να το παραδέχεται κιόλα, γιατί η Αιγυπτιακή κυβέρνηση ποτέ δεν έχει παραδεχθεί ότι υπάρχουν βασανισμοί. Όσον αφορά την παρατήρηση των εκλογών, αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Να σα υπενθυμίσω ότι υπήρξε και σχετική αίτηση, την οποία υπέγραψαν αρκετοί Αιγύπτιοι πολιτικοί, οι οποίοι ζητούν παρατηρητέ ε, στι εκλογέ, διότι δεν εμπιστεύονται την ε, ε, κυβερνητική διαχείριση τη εκλογική διαδικασία θα πρέπει να υπάρξει τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την μεταρρύθμιση και είναι θέμα πολιτικής βούληψης για τα ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουμε ότι απαφίεται σε εσά να παρακολουθήσετε και να τηρήσετε τις δεσμεύσεις οι οποίες δηλώθηκαν το 2003 όταν ε, ξεκίνησε η πολιτική ευρωπαϊκής γειτονίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα το απόγευμα στο Στρασβούργο, σε μια εβδομάδα δηλαδή, θα έχει την παρουσίαση της έκθεσης αυτής που θα προετοιμάσουμε αυτή και την παρουσίαση θα γίνει από τον Επίτροπο Φούλα που είναι υπεύθυνο για διεύρυνση. Ελπίζω λοιπόν ότι κάποια από τα μέλη μας θα είναι εκεί με όλες τις πληροφορίες που πήραμε σήμερα από τους ε, ε, ομιλητές εδώ. Σας ευχαριστώ για μια φορά που ήρθατε εδώ και προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. Τώρα, μπορώ να περάσω το τελευταίο πραγματικό σημείο τη μερικής διάταξης. Η πρώτη παρουσίαση της εχθές της Ευρωπαϊκή Ένωση για ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο υπό τους όρους της συνθήκης Λισαβόνας η ευθύνη για την έκθεση αυτή είναι στα χέρια της εκπροσώπου. Και ε, θα υπάρχει απογοήτευση που δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι αυτή είναι μόνο η απαρχή της ε, εξέτασης της έκθεσης αυτής εδώ στο Κοινοβούλιο. θα χαρείτε να μάθετε ότι θα υπάρχει παρουσίαση από την ίδια την είπατε εκπρόσωπο τον Ιούνιο στην Ολομέλεια. Και συμπίπτει με την έκθεση για τους πρόσπιστες των ανθρώπινων δικαιώματων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία ε, Αρνό από την Κομισιόν και τον κύριο Σιώκα που δεν είμαι σίγουρο το Συμβούλιο εκπροσωπεί με αυτήν την νέα δομή δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Χαίρομαι όμως πολύ που είσαστε εδώ. Κύριε Κύρκο θα αρχίσει από ό,τι κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και εμείς έχουμε εμπλεχτεί με αυτή την δομή όπως λέτε αλλά ελπίζουμε ότι θα βρεθεί η λύση. Παρουσιάζουμε την έκθεση αυτή μαζί με την ε, Διευθύντρια κυρία Βερονίκη Αρνό. Θα πρέπει να είμαι σύντομη βέβαια λόγω του προχειρημένου της ώρας. Θα σας δώσω με δύο λόγια μια εικόνα της έκθεσης αυτής γιατί διαφέρει όσον αφορά την μορφή της και ποιες είναι οι πρόσφατες εξελίξεις γεωγραφικά της νέας έκθεσης. Και μετά η Βερονίκη θα σας πει τα υπόλοιπα. Καταρχήν αυτό που προσπαθήσαμε να πετύχουμε την έκθεση αυτή ξέρετε πολύ καλά ότι θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή έχει σαν στόχο να αυξήσει την κατανόηση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό και ιδανικά θα γίνει η έκθεση αυτή ένα μέσο της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων αν αναγνωστεί αρκετά. Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε τους τομείς ε, αναχώρα της έκθεσης αυτής. Θα θυμόσαστε από παλιότερες εκθέσεις ότι ήταν πολύ τυχαίο ποιες χώρες καλύπταμε, πόσο τις καλύπταμε, πόσο αναλυτικά παρουσιάζουν τα στοιχεία. Τώρα όμως ε, έχουμε βελτιώσει κατόπιν πρωτοβουλίας ε, που πήραν η Σουηδική κυβέρνηση. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία και πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τι ε, εξωτερικέ πολιτικέ. Προσπαθούμε να είμαστε επίση πιο συστηματικοί, να αντικατοπτρίζουμε τη διαφορετική μορφή των κοινοτικών πολιτικών και να καταδείξουμε Πού μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Προσπαθούμε δηλαδή να βελτιώσουμε τα πράγματα επί τόπου. Θα σας πω τώρα γιατί είναι διαφορετική εκθέση αυτή και όσον αφορά τη μορφή με την οποία παρουσιάζεται. Πέρυσι το Σεπτέμβριο πάλι με Σουηδική Πρωτοβουλία η Επιτροπή Ασφαλείας του Συμβουλίου ε, αποφάσισε να ακολουθήσει κάποιες κατευθυντικές γραμμές για να αυξήσει την, οραματικότητα της, ε, την ορατότητα συγγνώμη, της ε, εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η έκθεση τώρα καλύπτει ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος, όχι από τον Ιούλιο στον Ιούνιο όπως παλιά. Κατ' εξαίρεση όμως επευθύνει μεταβατική έκθεση καλύπτει 18 μήνες. Δηλαδή 1η Ιουλίου 2008 έως 31 31η Δεκεμβρίου 2009. Αυτή είναι μια διαφορά. Υπάρχει διαφορά και στην μορφή, γιατί προσπαθήσαμε να είναι πιο ευανάγνωστο το κείμενο. Κάποιος που είδα πριν από τη συνεδρίαση μου είπε ότι αυτή τη φορά δεν την κούρασε το να διαβάζει την έκθεση αυτή ίσως κομπλιμέντων... Ναι, ότι πραγματικά βελτιώσαμε. Εμείς θέλουμε έκθεση αυτή τελικά να είναι ένα κείμενο που θέλουν οι αναγνώσεις μας να διαβάσουν. Και εξετάζουμε επίσης το θέμα των ε, μεταφράσεων του εγγράφου και κοιτάμε πώς θα μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε στα αραβικά, στα κινέζικα, στα φαρσί και στα ρώσικα και σε άλλες γλώσσες θα θέλαμε να το μεταφράσουμε αυτό το κείμενο της μελέτης. Επίσης δεν έχουμε δημοσιεύσει για πρώτη φορά αυτό το έγγραφο επί χάρτου, αλλά προετοιμάσαμε μια προσούρα που νομίζω ότι είναι πολύ ελκυστική, λεπτή ευανάγνωστη, για τους μη ειδικευμένου και η πλήρης έκθεση υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Και αυτό θα προωριστήσει και εκείνους που θέλουν να προστατεύσουν τα δέντρα, είμαι σίγουρη. Είναι πράσινη λοιπόν αυτή η έκθεση. Uh, um, uh, θα αναφερθώ τώρα στις ε, γεωγραφικές εξελίξεις και η Βερονίκ θα συνεχίσει μετά. Όσον αφορά την πολιτική, αυξήσαμε τον αριθμό των διαλόγων και διαβουλεύσεων και συζητήσεων για ανθρώπινα δικαιώματα που είχαμε με τρίτες χώρες. Έχουμε 40 περίπου αυτή τη στιγμή. Ήδη βρισκόμαστε στο τρίτο γύρο με κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας με τι οποίε είχαμε ξεκινήσει στο Ισπικστάν παραδείγματο χάρη, είχαμε στο τέταρτο γύρο, ξεκινήσαμε νέου διαλόγους με διάφορες χώρες, όπως με την Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Λευκορωσία, Ινδονησία. Ξεκινήσαμε επίσης υβριδικού διαλόγους με χώρες Λατινικής Αμερικής, δηλαδή και στη Νέα Υόρκη και εδώ, κάναμε μια σοβαρή επανεξέταση του διαλόγου με την Κίνα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Η ανατολική εταιρική σχέση ξεκίνησε επίσης με την τελευταία, μετά την τελευταία έκθεση και η Ένωση για τη Μεσόγειο. Ε, ξεκινάμε να εξετάσουμε τα θέματα αυτά με τους δικούς απεσταλμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζω ποια είναι τα κέρια θέματα. Είχαμε μία προσπάθεια mainstreaming τον Γενάρη που ήταν πολύ επιτυχής. Τώρα προχωράμε στη διαχείριση της κρίσης ε, σε αποστολές ε, και εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα που είναι η αποστολή στην Γεωργία όπου υπήρχαν σημαντικά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μιας αρχής. Θα σταματήσω αυτό και θα δώσω το μικρόφωνο στη Βερονίκ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς το ίδιο κάναμε όσον αφορά την κατάρτιση για τις ε, επιχειρήσεις ε, αμάχων ε, είναι γεγονός όμως ότι εκτός από τη διάκριση μεταξύ αμάχων και στρατιωτικών πρέπει να υπάρχει και αυτή η πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά τώρα τον, ε, ε διπλωμα, τις διπλωματικές αποστολές που έχουμε τώρα επί τόπου, ε, έχουμε περίπου... Ε, 200 που έχουν focal points και εκεί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ενημέρωση που είναι αρκετά ε, ενεργός ε, όχι μόνο στα focal points, ε, όχι μόνο στα focal points αλλά και με τους πολιτικού σε τοπικό επίπεδο για να συμμετέχουν περισσότερο και οι πολίτες. Οι οκτώ κατευθυντήριες γραμμές όλες αναθεωρήθηκαν ε, από το 2008. Εγκρίναμε και νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη βία κατά των γυναικών που είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τώρα την συνοχή μεταξύ των ε, πολυμερών και διμερών ε, ζητημάτων. Ε, σας μίλησε η Ρίνα για 40 διαλόγους και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να συνδέσουμε το διμερές με το πολυμερές και είναι κάτι το οποίο αναφερόταν και στην έκθεση της κυρίας Αντρικέινε για τις εργασίες στην Γενέβη. Όσον αφορά τώρα τη Γενέβη την ίδια, ήμασταν πολύ πιο δραστήριοι στη συμμετοχή μας, στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίξαμε και ελπίζω να ήταν ορατό αυτό στη διαδικασία του ε, UPR. Και επίσης ε, προσπαθήσαμε να έχουμε περισσότερες επαφές με τις τρίτες χώρες ε, στο πλαίσιο των διαφόρων, προετοιμασιών για τη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όσον αφορά την προετοιμασία της αναθεώρησης ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2011, λάβαμε υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την εφαρμογή, υπάρχει ένα μέσο ε, Τη δημοκρατία δημοκρατίας ε, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περίοδο αναφοράς κάθε φορά που μπορέσαμε να εφαρμόσουμε, να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό έχουμε 238 εκατομμύρια για 900 προγράμματα σε 100 χώρες. Αυτό σημαίνει πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις σε πολλές χώρες, κυρίως χώρες ΑΚΕ, αλλά και στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις τοπικές επίσης. Είναι λοιπόν κάτι το πολύ σημαντικό το να έχουμε τέτοιου είδους μέσο που λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και όσον αφορά τώρα τις θεματικές ενότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρά το γεγονός ε, ότι σας είπε η Πρόεδρος στην αρχή της σημερινής ε, συνεδρίασης ε, κάποια αρνητικά αποτελέσματα υπάρχουν αρκετές χώρες, όλο και περισσότερες που είτε αναστέλουν τη θανατική καταδίκη είτε σιγά σιγά την καταργούν 106 χώρες το 2008 προσχώρησαν στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών κατά τη θανατική καταδίκης και ελπίζουμε φέτος, επειδή έχουν περάσει δύο χρόνια, να έχουμε ακόμη περισσότερες χώρε που θα μας υποστηρίξουν σε αυτό. Κάτι ακόμη το οποίο είναι επίση αρκετά θετικό είναι ο αυξανόμενος αριθμός των χωρών, μεταξύ των οποίων και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι συμβαλόμενα μέρη ή έχουν επικυρώσει το επιπρόσθετο πρωτόκολλο τη σύμβασης ε, ε, για το βασανισμό. Αυτά ήθελα να πω σε σχέση με την πρόοδο της εξελίξης ε, από την τελευταία έκθεση. Οπότε, σε επίπεδο πολυμερές, ε, πολλή εστίαση στις δραστηριότητες στην Γενέβη, στο outreach, όπως επίσης και στο διάλογο, ε, στη σχέση μεταξύ διμερούς και πολυμερούς διαλόγου ενίσχυση και ενημέρωση όλων των κατευθυντηρίων γραμμών που είναι η πολιτική μας βίβλος ουσιαστικά, εφαρμογή αρκετά ενεργώς ε, του Μηχανισμού για τη Δημοκρατία και τα ε, Ανθρώπινα Δικαιώματα, πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και βεβαίως ε, μια ευρύτερη θεώρηση ε, της, του βασανισμού και της θανατικής καταδίκης. Τώρα, ποιες είναι οι προοπτικές για την επερχόμενη περίοδο. Μιλήσατε, κυρία Πρόεδρε, ε, για τις ε, ελπίδες ε, ε, που έχετε να αποθέσει στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης αναφερθήκατε στις αξίες που είναι θεμελιώδης πυλώνας και αναφερθήκατε επίσης και στο συνδυασμό των διαφόρων μέσων η χάρτα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι επίσης κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και θα δούμε πώς θα γίνει να αποτελεί υποχρέωση προκειμένου να έχει ένα πιο απτό αποτέλεσμα και επίσης πώς θα αρχίσουμε να ε, προετοιμάζουμε την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της ε, Ευρώπης. Ε, βέβαια και το δικαστήριο θα έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ενισχυμένο ρόλο για τα ζητήματα τα εξωτερικά και βέβαια και στα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι τμήμα αυτού του τομέα. Έχουμε και μία αντιπρόεδρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό δίνει μεγαλύτερη αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον ε, τρίτο ε, πυλώνα και νομίζω ότι η ανάπτυξη του, προγραμμάτου, του προγράμματος της Στοκχόλμης και κυρίως για την εξωτερική πτυχή είναι κάτι το οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο. Τώρα, οι προκλήσει το γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, πρέπει να είμαστε συνεκτικοί, να υπάρχει συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων και να είμαστε και αρκετά αξιόπιστοι προς τα έξι. Νομίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει πολλές τέτοιες δυνατότητες, αλλά πρέπει το κάθε πράγμα να έχει τη ε, θέση του και το, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι κάτι που θα αρχίσει να λειτουργεί με πιο ορατό τρόπο πρέπει να υπάρχει, πρέπει και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ό,τι κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι επίση πιο απτά, πιο ορατά. Είπατε κι εσείς ότι Είπατε και εσείς ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ε, ε, σχετικά με την γεωγραφική κατανομή ε, και τη γεωγραφική εκπροσώπηση και είπατε ότι ανησυχούν κάποιοι ευρωβουλευτές για το θέμα αυτό. Βεβαίως το λάβαμε υπόψη. Όσον αφορά τώρα την Βελγική Προεδρία που είναι πολύ σημαντική γιατί εκεί θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ειδικότερα όσον αφορά τις πολυμερείς συζητήσεις και τη σημασία του ρόλου της Προεδρίας στην εξωτερική εκπροσώπηση. Συνεργαζόμαστε με την επερχόμενη Βελγική Προεδρία για να υπάρξει ένα πρόγραμμα εργασία όταν λέω εμείς εννοώ εννοούμε η κοινή εκπροσώπηση, εγώ και η συνάδελφος, ε, θα υπάρξει και συνάντηση πολύ σημαντική, ένα φόρουμ με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που Βελγική Προεδρία θα συζητήσει ακριβώς όλα αυτά τα ζητήματα εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ε, συνοχή εσωτερικών και εξωτερικών ε, δράσεων και επίσης πτυχές της εξωτερικής πολιτικής που είναι πολύ σημαντικές σήμερα γιατί έχουμε τα 10 χρόνια ε, την σύσταση 1325 τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη. Επίσης η αναθεώρηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2011. Όλα αυτά λοιπόν είναι ήδη πολλά και υπάρχει βέβαια και όλα αυτά θα συζητηθούν στις 12 και 13 Ιουλίου στο Φόρουμ για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις υπό Βελγική Προεδρία. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια μεταβατική περίοδο που καθιστά ε, τις διαδικασίες λίγο πιο δύσκολες μερικές φορές και είναι πολύ σημαντικό ε, να συνεργαστούν όλα τα ευρωπαϊκά όργανα ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις δύο παρουσιάσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι μπορούμε μέσω αυτής της εκθέσεως να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές μας θέσει και σημειώνω επίσης το γεγονός ότι μας δίνεται ήδη η δυνατότητα να συζητήσουμε τις νέες περιόδους, διότι η περίοδος που καλύπτει αυτή η έκθεση είναι προς το τέλος Ξεκίνησε και η εφαρμογή της ε, συνθήκης Λισαβόνα το Δεκέμβριο του 2009, οπότε ελπίζω να έχουμε και κάποιες αλλαγές ε, θετικές. Να δώσω πρώτα το λόγο στους ε, αντιπροέδρους, την κυρία Ανρική. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Είχαμε πολύ σημαντικές απαντήσεις από πλευράς Κοινοβουλίου στην προηγούμενη έκθεση. Και η τελευταία έκθεση του Κοινοβουλίου που ετοίμασε ο κύριο Ομπιό ε, ζητά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να έχει συγκεκριμένους ποσοτικοποιημένους δείκτες προκειμένου να ε, μπορούμε να μετρήσουμε και την αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής. Ε, να δούμε δηλαδή κατά πόσο γίνεται κάτι τέτοιο. Σημειώνουμε επίση ότι ο τίτλο πλέον περιλαμβάνει και τον όρο «Δημοκρατία», γεγονό που αντικατοπτρίζει τα σημαντικά αποτελέσματα που είχαμε το φθινόπωρο για τα θέματα της δημοκρατίας και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να περιμένουμε και την επόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της δημοκρατίας, κάτι βέβαια το οποίο είναι ξεχωριστό από αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το Κοινοβούλιο επίσης ζήτησε να γίνει σύγκριση μεταξύ των ε, διαφόρων διαλόγων και διαβουλεύσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φαίνεται να μην είναι τόσο εύκολο σε αυτή την έκθεση να γίνει σύγκριση. Θα δούμε κατά πόσο να απαιτείται κάτι τέτοιο. Έχω την αίσθηση ότι τους τελευταίους μήνες, ε, όπως και εσείς μάλλον, αλλά φαίνεται ότι διαπιστώνουμε ότι παρά το διάλογο και τις διαβουλεύσεις τα πράγματα είναι απογοητευτικά και μένουν αρνητικά. Και θα πρέπει ίσως να δούμε μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό επί του θέματος. Μία ακόμα παρατήρηση ίσως που θα μπορούσα να κάνω. δεν δίνονται πολλά στοιχεία σε αυτή την ετήσια έκθεση για την ε, πρόοδο αναχώρα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ίσως θα πρέπει να τα δούμε και αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Αρκίνε, η οποία μπορεί και να είναι και η συγγήτρια από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, αντίστοιχη έκθεση, θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω λιθανικά σήμερα. να σας πω ότι είχα ένα ραντεβού με τον οδοντίατρο και μου είναι λίγο δύσκολο να προσπαθήσω να μιλήσω ξένη γλώσσα σήμερα. Γι' αυτό θα μιλήσω λιθουανικά. Να σας πω ότι περιμέναμε με ανυπομονησία την έκθεση αυτή και εκτιμούμε το γεγονός ότι μπορούμε να ακούσουμε την έκθεση αυτή εδώ σήμερα στην υποεπιτροπή μας. Ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σταθώ σε κάποια σημεία, να επισημάνω ότι δεν είναι πρόθεσή μου να μειώσω τη σημασία της έκθεσης αυτής. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες πτυχές οι οποίες δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως και θα ήθελα να σταθώ σε αυτές. Η κυρία Χαουτάλα ήδη ανέφερε κάποια στοιχεία ε, και θα ήθελα να πω κι εγώ ότι αν δείτε τα σχετικά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και, για και ψηφίσματα τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, έχουμε ζητήσει επανειλημμένους από το Συμβούλιο να έχει ποσοτικοποιημένους στόχους, ε, κριτήρια για τις χώρες ε, και για τα οριζόντια ζητήματα που τις αφορούν και να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι που προσπαθεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε στο τέλο του έτου, όταν κάνουμε τον απολογισμό μα, να βλέπουμε κατά πόσον ήταν αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσον υπήρχαν ε, στοιχεία, ποσοτικοποιημένα στοιχεία. Οι πολίτε που διαβάζουν τις εκθέσεις αυτές περιμένουν απαντήσει σε πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει, κατά πόσον η κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει βελτιωθεί στους τελευταίους 12 μήνες και κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρεσβεύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της, έχει επιτύχει τους στόχους της και κατά πόσον έχουν δαπανηθεί τα χρήματα των φορολογουμένων με αποδοτικό τρόπο. Διέτρεξα λίγο την έκθεση που συζητάμε σήμερα και νομίζω ότι αυτή η διάσταση δεν συμπεριλαμβάνεται. Δεν υπάρχει αυτή η πτυχή της αξιολόγησης. Αν διαβάσω σε μια έκθεση ότι η κυβέρνηση μια συγκεκριμένη χώρα έλαβε εκατοντάδε αιτήσει για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, θα ήθελα να γνωρίζω και ε, ποια υπήρξε η συνέχεια, τι αποτελέσματα είχαμε. ο εξορθολογισμός των ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, στις ε, Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας υπενθυμίσω ότι στη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας το 2008 υπήρχε μια πρόταση επί του θέματος και διαβάζοντας την έκθεση αυτή θα ήθελα να μπορούσα να διαπιστώσω τι ε, αποτελέσματα είχαμε στο συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχει μια σελίδα για τη Ρωσία η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες και λέει ότι συζητήθηκαν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία. Αντίστοιχα όμως στοιχεία δεν έχω στην κατάσταση της Κίνας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς έχει η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται τα ίδια φαινόμενα. Κατόπιν, διάλογος και διαβουλεύσεις ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έκθεση του 2008 περιείχε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για το θέμα αυτό και ήταν πολύ εύκολο να γίνει η σύγκριση ε, μεταξύ της προόδου που επετεύχθη τώρα και στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή η δομή της έκθεσης είναι διαφορετική και αυτή η ανάλυση είναι πολύ πιο δύσκολη. Έχω την εξής ερώτηση λοιπόν. τι γίνεται με το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ξέρω ότι υπάρχουν τέσσερις ε, δομές για το διάλογο σε ανθρώπινα δικαιώματα. Διαρθρωμένος διάλογος, ε, τοπικός διάλογος, διάλογος ο οποίος γίνεται σε συγκεκριμένε υποεπιτροπές και διαβουλεύσεις για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αργεντινή, Κολομβία, Βραζιλία, Χιλή. Γίνονται διαβουλεύσεις χρησιμοποιώντας αυτή την, ε, το επίπεδο το τοπικό, σε επίπεδο τοπικών εκπροσώπων. Και φυσικά γνωρίζω ότι οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνε για το διάλογο αυτό στις χώρες αυτές. Ξέρω ότι οι ευρωβουλευτές δεν έχουν πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία ε, απεικονίζουν την πορεία του διαλόγου. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τι θα πρέπει να περιμένουμε. Τι θα πρέπει να περιμένουμε όταν θα ξεκινήσει και τις εργασίες της η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι χρήζει της ε, προσοχής μας, ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή φόρα. Οι κυρίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Κάοκα και η κυρία Αρνό, αναφέρθηκαν σε αυτά, αναφέρθηκαν και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο ρόλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένος η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας ε, έχει παραστεί σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου αυτού τέσσερις φορές και πολλές φορές έχουμε αντιπροσωπείες ε, στην, ε, στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Και φαίνεται σαφώς ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις και μάλιστα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα είναι εμφανή και αυτή η κατάσταση φυσικά είναι προς όφελος των αντιπάλων μας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις και για το συγκεκριμένο θέμα. κάτι επιπλέον. Η κατάσταση σε κάθε χώρα. Κατανοώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια έκθεση να περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για μια χώρα. Παρ' όλα αυτά, κάποιες σημαντικές πτυχές θεωρώ ότι έχουν παραλυφθεί. Ας δούμε επί παραδείγματι την Κίνα. Ξέρω ότι στη διάρκεια του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα είχαμε την εκτέλεση ενός ε, αυστριακού πολίτη ε, λόγω εφαρμογής της θανατικής καταδίκης. Ε, άλλο παράδειγμα, ένας Βρετανός πολίτης εκτελέστηκε επίσης γιατί του είχε επιβληθεί η θανατική ποινή. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται σε μια έκθεση αυτού του τύπου. Στη Δημοκρατία του Κονγκό Η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ε, έχει ενεργό ρόλο στις ε, δραστηριότητες του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά αρνείται να εφαρμόσει οποιαδήποτε απόφαση έχει εκδοθεί για την ε, χώρα της. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να εκφράσω μια επιθυμία μου. Θα ήθελα οι συνάδελφοι στην Υποεπιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να γνωρίζουν ότι αυτή η ετήσια έκθεση είναι μία από τις πιο σημαντικές, αν όχι η πιο σημαντική έκθεση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, προώθηση της δημοκρατίας ανά τον κόσμο και ελπίζω η έκθεση αυτή να λάβει και τη δέουσα προσοχή και να έχουμε και αρκετά σχόλια. Όταν αναφερθήκατε για την Κορέα, εγώ άκουσα Αλλά εννοούσατε εσεί Βόρειο Κορέα. Α, εντάξει. Η Μπάρμπαρα Λόχπιλ έχει το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση. Είναι πάρα πολύ καλό να δει κανένα πόσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Λάκα είπε επίση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντάξει κανένα μια τέτοια έκθεση. Αναρωτήθηκα, για ποιον έχει γραφεί αυτό. Αν κανένα είναι ε, ειδικό ή ενδιαφέρεται για κάποια χώρα, δεν ενδιαφέρεται για τα, τις άλλες χώρες. Λοιπόν, εάν ο στόχος είναι να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον, ε, έχω κάποιες ιδέες. Βέβαια, δεν υπάρχει ένας ιδανικός τρόπος για να γράψει κανένας μια τόσο ογκώδη έκθεση, αλλά θα μπορούσατε ίσως να ξανασκεφτείτε Ίσως ήταν καλό κάθε έκθεση να έχει ένα κύριο θέμα, κάπως όπως είναι και η έκθεση του Κοινοβουλίου. Και εκεί να περάσετε πραγματικά ε, εις βάθος της ανάλυσης. Ένα θέμα είναι καλύτερο από το κάθε χώρα. Να δείτε δηλαδή ποια είναι τα κοινοτικά μέσα που οδήγησαν σε επιτυχία. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να δει κανένα πόσο δύσκολο είναι να πετύχει ε, πρόοδο στην εφαρμογή και να δείξετε πού υπάρχει πρόβλημα και πού δεν έχει υπάρξει πρόοδος. Αυτό νομίζω θα κινητοποιήσει περισσότερο το ενδιαφέρον. Θα κάνει το πρόβλημα πιο κατανοητό, γιατί αλλιώς η έκθεση είναι πολύ στεγνή θα έλεγα. Στις αρχές της έκθεσης αναφέρονται διάφορα θέματα καθώς επίσης και θέματα συνοχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω αυτά που λέγονται εκεί, ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αυτοκριτική. Είναι ενδιαφέρον να δούμε την ε, κριτική σε κάθε στάδιο και είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η αντίρρηση Ευρωπαϊκή Ένωσης εκείνου που επικρίνουν τη στάση του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν έχουμε περισσότερες ε, συστάσει από την UPR προς ευρωπαϊκές ε, χώρες, θα πρέπει να κάνουμε μια συλλογή, να δούμε ποια είναι τα πιο συχνά ε, επεισόδια παραβασης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ένα θέμα τρομοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Σημείο 9. Δεν αναφέρεται καμία αυτοκριτική όσον αφορά τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και στην αρχή μιας αυτοκριτικής θα πρέπει νομίζω κάτι εδώ να αναφέρεται. Είναι καλό να γκομιάζουμε τη ΣΥΠΑ που έκλεισα τον Γκαντάναμο. Αλλά αν δεν αναφέρεται τίποτα για την Ευρώπη, ε, εμένα δεν με αρέσει καθόλου αυτό. Και θα πρέπει να επικρίνουμε επίση κάποιε διατυπώσει που υπάρχουν. Σελίδα 74, παραδείγματο χάρη του εγγράφου που προετοιμάστηκε για δική μα επιτροπή λέει ξεκάθαρα ότι χρησιμοποιείται βασανιστήρια στο Κουαντάναμο. Αλλά κατά τα άλλα στην παράγραφο δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο. Αναφέρονται για σκληρές μεθόδους με μέθοδοι ανάκρισης. Γιατί όταν υπάρχει βασανισμός θα πρέπει να τον λέμε. Να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν επιτρέπεται. Μετά λέτε ότι προετοιμάστε για την σύνοδο των 20, την G20, που θα πρέπει να έχει μια πιο ευρεία ανθρώπινη διάσταση. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η ουσία αυτή τη ανθρώπινη διάσταση για την επόμενη G20. Και λέτε επίσης ότι σε σχέση με την ανάπτυξη και την κοινωνία των πολιτών Στη 36 αναφέρομαι τώρα. Θα πρέπει να συζητηθεί περισσότερο με οργανώσει τη κοινωνίας των πολιτών ποιες είναι οι κύριες ε, προκλήσεις για τη συμμετοχή της κοινωνία των ε, πολιτών στην εφαρμογή τη αναπτυσσιακής βοήθεια. Και αναφέρεται εδώ στο ειδικό έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί για το 2010. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν αυτό να το ακούσω. Και επίση λέτε ότι η Κομισιό ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2009 μία μελέτη για το νομικό πλαίσιο του ανθρώπινου δικαιωμάτων και περιβάλλοντο. Και αυτό θα με ενδιαφέρει να ακούσω τι λεπτομέρειε να ξέρω πόσο έχει προχωρήσει. Γενικά πάντως είναι ένα έγγραφο που πραγματικά θα διευκολύνει πάρα πολύ την εργασία μα. Αλλά για να επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, αν θέλετε να το διαβάσουμε το έγγραφο αυτό που δεν έχουμε τις λεπτομερείς πληροφορίες, θα πρέπει να είναι περισσότερο κίνητρο για σκέψη. Ναι, αυτό ήταν πραγματικά και η γραμμή σε εμά που εισαγάγαμε την έκθεση αυτή. Υπήρχαν βέβαια πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλά σχόλια και δεν έχουμε σχόλ, χρόνο για να απαντήσετε. Μήπως μπορείτε να έχετε μια πολύ σύντομη παρέμβαση τώρα και να επανέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα στο μέλλον γιατί η παρουσίαση θα γίνει στην Ολομέλεια, η Επιτροπή θα προετοιμάσει τη δική της έκθεση. Η αρχή είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή τη συζήτηση. Αλλά πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα την ειλικρίνεια και το ανοιχτό πνεύμα συνεργασία που έδειξε η Κομισιόν. Αυτό θα μα βοηθήσει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ελπίζω να μην θεωρήσετε αγενή, αλλά θα σας ζητήσω να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι. για να έχουμε και δύο λόγια για τη διαβούλευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Τρία λεπτά λοιπόν θα έχουμε γι' αυτό. Προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη, αλλά δεν θα απαντήσω όλα τα ερωτήματα τότε. Ναι, το καταλαβαίνω. Ίσως δεν χρειάζεται αυτή τη φορά να τα απαντήσετε όλα. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε αυτά που μου έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση όσον αφορά τους ποσοτικοποιημένους στόχους και αποστολές. Δεν είναι όλα ποσοτικοποιήσιμα. Δεύτερον, Όσο και να θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι δράσει Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζουν τόπου τα πράγματα, δεν ισχύει πάντοτε αυτό. Δεν ισχύει επίσης πάντοτε ότι αν υπάρχει αλλαγή προέρχεται από τη δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει, Ένωσης. πρέπει να είμαστε ε, πάρα πολύ ειλικρινεί ω προ αυτό, παρά το γεγονό ότι μπορεί να μα αρέσει. Και αυτό βέβαια πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη όταν έχουμε να κάνουμε με αξιολόγηση διαλόγων. Ε, πόσο δηλαδή αποδίδεται η αλλαγή επιτόπου στη συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι όμως πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή πολύ ευρύτερα. Λαμβάνουμε όμω υπόψη το σχόλιο. Όσον αφορά τώρα τα διάφορα είδη διαλόγων και διαβουλεύσεων. Ναι, τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες υφίστανται, τις αναφέρατε κι εσεί, αλλά αποφασίσαμε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι όσον αφορά τη Λατινική Αμερική θα υπάρχει ένας ε, υβριδικός διάλογος ε, διάλογο σε τοπικό επίπεδο με λίγο διαφορετική προσέγγιση για το Μεξικό αλλά θα υπάρχει και πρόσβαση των διεθνών ε, φόρα για παράδειγμα στην Νέα Υόρκη ή στη Ουάσιγκτον για τα διεθνή φόρα και το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις στη Γενέβη και στη Νέα Υόρκη, έχουν διαφορετικές απόψεις και εδώ. Σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Λόχ Μπίλερ. Η πρότασή σας, ε, μια θεματική ενότητα αναέκθεση είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πραγματικά, ε, αξίζει τον κόπο, πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε. και να ακούσουμε τα κράτη-μέλη που όντω έχουν κάτι να ε, συνεισφέρουν. Τώρα, περισσότερη εστίαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα ο στόχο είναι να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα εξωτερικά ζητήματα. Δεχόμαστε την κριτική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι σε θέση να μιλά για ανθρώπινα δικαιώματα σε άλλες χώρες μόνο αν ε, ε, μιλούμε και για το τι συμβαίνει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομίζω ότι θα έπρεπε να το εξακολουθήσουμε να το συμπεριλαμβάνουμε στην έκθεση. Καλύτερα να σταματήσω επειδή μου είπατε να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά. Μπορούμε να την κάνουμε χωρί διερμηνία. Ευχαριστώ του διερμηνείς οι Πρόεδρου. Oh, thank you very much, Heidi. I just wanted to say that uh, the nature of the beast, it's difficult